Αλλά ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με πολύ λίγα μέλη της Επιτροπής. Βλέπω τον κύριο Γιάρ που δεν ήταν το πρωί. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο σημείο 12. Όχι, στο σημείο 13 διορθώνει η πρόεδρος. Σας το συγγνώμη. Το 13 as were postponed because we, we don't take them now. We go on to the. Oh, I didn't know that. Uh, postponed for the next. I thought for the afternoon. So I thought that uh, number 20. Λοιπόν, είχα την εντύπωση ότι το 12 θα το συζητούσαμε τώρα το απόγευμα, αλλά ξεκινάμε το 13. Το οποίο αφορά διακριτική μεταχείριση. του Lord ε, Richard Inglewood. Είναι συγκεκριμένη αναφορά. Δεν είναι. Το, το αξίωμα των Λόρδων ε, και συζητάει για το αν θα έπρεπε να ε, το χάνει κανείς εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι εδώ από τη μεριά της Επιτροπής ο κύριος Βάση. Βάση, ο Τίμπορ Βάση, παρακαλώ. Είναι έτοιμος να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ. Oh, please do. Start. Είμαστε στο 13. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για που μου δώσατε το λόγο. Κοιτάξτε, αυτή η αναφορά αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα της Βρετανικής νομοθεσίας και αφορά την δυνατότητα ε, των κληρονόμων να, να, πάρουν, να πάρουν την έδρα τους αν, ελεγχθούν, ε, ε, αν εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 76. Όσον αφορά ε, την εκλογή, το, το νόμο για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία, το 2002 με την, με την απόφαση 772 καθορίζονται οι περιπτώσεις ασυμβίβαστου και προβλέπεται ανάμεσα στα άλλα ότι το αξίωμα μέλους του Εθνικού Κοινοβουλίου είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το σύστημα και ο νόμος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος ε, λόγω των ε, παραδόσεων. Τα μέλη του Κοινοβουλίου, τα Βρετανικά μέλη του Κοινοβουλίου, ε, παρετούνται από το εθνικό τους αξίωμα αν εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφύγουν τη διπλή θητεία. Όμως μέλη ε, της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ε, ελάβει το αξίωμα ε, ως κληρονομικό δικαίωμα δεν μπορούν να παρατηθούν και σόβιο δικαίωμα δεν μπορούν να παρατηθούν. Γιατί όπως σας είπα είναι ισόβια μέλη της Βουλής των Λόρδων. Όμως για να, μπορέσουμε να για να μπορέσει να υπάρξει ευθυγράμμιση της, ε, της, της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την πράξη του 1976 για την εκλογή ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεκρίθησε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2008 μια νομοθεσία, ε, ένας κανονισμός μάλλον, που προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής Τη ιδιότητα του μέλου της Βουλής ε, του Λόρδου στην περίπτωση που έχουμε ισόβια μέλη. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο αναφέρεται στην αναφορά έχει να κάνει με το εξή. Αυτός ο κανονισμός δεν αναφέρει την, οδηγία, τη δυνατότητα αυτή αναστολής ενώ την αναφέρει στα ισόβια μέλη, δεν την αναφέρει ε, στα μέλη ε, κληρονομικό δικαίου. Άρα λοιπόν, ε, εμείς κάνα, έγινε μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδε στην περίπτωση αυτών των hereditary peers που εκλέγονται ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. για το πώ μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντά του ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη αυτά, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολή του αξιώματό του και τη ιδιότητά του ω μέλου τη Βουλή των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι ε, είδε ότι εδώ υπάρχει περίπτωση ασυμβίβαστου ε, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Οκτώβριο του 2009 απέστειλε επιστολή στις Βρετανικές Αρχές όπου εξηγούσε, ανέπτυσε αυτές τις ανησυχίες και ζητούσε από τις Βρετανικές αρχές να ε, κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Απεστάλλει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία επιστολή στην Βρετανική μόνιμη αντιπροσωπεία τον Οκτώβριο του 2009. Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει τίποτα στο μεταξύχρονικό διάστημα, δεν πήραμε την απάντηση από τις Βρετανικές αρχές και σήμερα είμαστε σε επαφή μαζί τους και ζητάμε την απάντησή τους. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. I'm, I'm really here just... Κυρία Λάτφορντ, Κοιτάξτε, έχω ενδιαφέρον για το ζήτημα, γιατί εμπίπτω στην κατηγορία που ωφελήθηκε από τον κανονισμό αναστολής του 2008. Είμαι ισόβιο μέλος ε, στη Βουλή των Λόρδων και μπόρεσα να ωφεληθώ από την προσωρινή αναστολή ε, που μου επέτρεψε να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ήξερα ότι δεν προβλέπεται το ίδιο για τα κληρονομικά μέλη, Βεβαίω καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα απερχιωμένο ο θεσμό ε, ο θεσμός η Βουλή των Λόρδων. Δεν χρειάζεται να σα πω πολλά για το ζήτημα αυτό. Τώρα, τι να, ε, τι να σα πω. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το, το ζήτημα και θέλω να δω τι εξηγήσει θα δώσει η Βρετανική κυβέρνηση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική επιστολή. Πάντω σίγουρα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες των μελών ε, της Βουλής των Λόρδων. Και υπάρχει διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά το, την δυνατότητά του να αναλάβουν καθήκοντα στο, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση 2002 του Συμβουλίου. Δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε μπορώ να κάνω ένα σχόλιο αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω ότι με ενδιαφέρει το ζήτημα και είμαι εδώ για λόγους ε, ενδιαφέροντος προσωπικού αλλά και ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λάτφορτ. Ε, ο κύριος Λό θα ήθελε να συμβάλλει στη συζήτηση. Um, members, this item was... Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό ε, ήρθε στην ημερήσια διάταξη μετά από αίτημα του σε Ρόμπερτ Άτκιν και μετά από μια συζήτηση στην προηγούμενη επιτροπή. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας... Ε, στο, στη γνωμοδότηση που έχετε από την Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, Θεσμικών Υποθέσεων, που εδόθη ακριβώς πριν από τις ε, τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. Στο μεταξύ χρονικό διάστημα η Γραμματεία πήρε άτυπες ανακοινώσεις με τη μορφή ηλεκτρονικού, μηνυμάτου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου και ως αποτέλεσμα η κυρία Ματσόνης, η πρόεδρος, απέστειλε ε, επίσημη επιστολή για άλλη μια φορά στις, Ηνωμένες, ε, αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας επίσημη απάντηση ε, στο, στην αναφορά του Λόρδου Ίγκλιγουτ. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε συγκεκριμένο ζήτησε συγκεκριμένα ο Σε Ρόμπερτ να ενταχθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Καταγράφεται στα πρακτικά ότι αναφέρθηκε το ζήτημα και ότι θα επιστρέψει μόλι θα έχουμε την την επίσημη ε, τοποθέτηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό το στάδιο, από σας είπα, μέσα από την άτυπη επικοινωνία μου μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ε, κατάλαβα ότι εξετάζεται το ζήτημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από ό,τι κατάλαβα και από το ε, Υπουργικό Συμβούλιο και από το Γραφείο του Πρωθυπουργού και φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχουμε μια απάντηση. Και φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα θα πάρει απάντηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. For, uh, Λοιπόν, ωραία. Περιμένουμε την απάντηση από τις Βρετανικές Αρχές και πάμε στο 14. Uh, uh, λοιπόν, ο αναφέρον θα παρουσιάσει το θέμα. Yeah, sit down here. And you have to speak here. You are going to be more comfortable. So, okay. Chairperson, um, committee. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, χαίρομαι που κρίνετε παραδεκτή την αναφορά και μας επιτρέψατε να την παρουσιάσουμε. Εμείς είμαστε στο νότο της Ιρλανδίας, βλέπετε και στον χάρτη. 15 χιλιόμετρα βόρεια του Κόρκ ε, λέγομαι Μπάρι Κάρτιν και εκπροσωπώ μια κοινοτική εταιρεία. Είμαστε κατά της λειτουργίας λατομείου. Η εταιρεία λέγεται John ε, A. Woods Limited και έχει ε, γίνει και προσφυγή. Η αναφορά μας θέλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κοινοτικές ε, οδηγίες και την νομοθεσία γενικότερα σε σχέση με το πόσιμο νερό μεταξύ άλλων. Ε, παραβιάζονται ε, η οδηγία για τα ύδατα και η οδηγία για τις ΕΠΕ, επιπτώσεις περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Βλέπετε εδώ την ε, λειτουργία ε, του λατομείου αυτού και η δράση του και στον υδροφόρο ορίζοντα. Γιατί έχουν κάνει λατόμηση μέχρι το έδαφος του βράχου κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Οπότε επηρεάζεται ο υδροφόρος ορίζοντας που ε, δεν είναι πολύ, σε πολύ μεγάλο βάθος, είναι κάτω από ένα λόφο. Αυτός ο υδροφόρος ορίζοντ ε, εδώ και 1200 χρόνια λειτουργεί. Ε, προσφύγαμε στις ε, τοπικές αρχές και τους είπαμε για το πρόβλημα, δηλαδή ότι το λατομείο με τις λειτουργίες του μειώνει τα υδάτινα αποθέματα και απαλήφει το φίλτρο που υπάρχει ως προστασία στον υδροφόρο ορίζοντα. Βλέπετε ότι ο, ο χώρος της λατόμησης βρίσκεται ε, μέσα σε αυτόν τον δακτύλιο που συμπεριλαμβάνει και τις ε, ε, πηγές του ύδατος και το υδροφόρο ορίζοντα. Το 1974 ε, είχε δοθεί έκταση για 5 εκτάρια ε, λατόμηση στην εταιρεία. Βλέπετε, μόνο 5 εκτάρια είναι σκιασμένη περιοχή. Και μετά το 90, όχι το 89 με συγχωρείτε, ο υπεύθυνος του σχεδιασμού ε, πήρε την εντολή να μην ανανεώσει την άδεια. Ενημερώθηκε για την λήξη. Τέσσερες ιδεολογικές αξιολογήσεις έγιναν ε, και μία από την ίδια την κοινότητα και μία από τον υπεύθυνο του Λατομείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο μελέτες συμφωνούν ότι ο υδροφόρος αυτός ορίζων είναι ιδιαίτερα ευάλωτος. Επίσης ε, εδώ στο slide καταγράφουμε τη συνολική περιοχή που ξεπερνά τα 40 εκτάρια. το νερό έρχεται στην περιοχή και περνάει από το σύστημα προς ε, την πηγή που βρίσκεται εδώ 600 ε, μέτρα από το λατομείο. Είναι επίσης ε, και για την περιφέρεια σημαντικός ο υδροφόρος ορίζων γιατί πάνω από 50.000 άνθρωποι καλύπτονται από εκεί προς τον Νότον σε πολλές πόλεις και στο νότο της, ε, του Κόρκ. Ε, τρεις ποταμών ε, περνούν από εδώ. Το νερό λοιπόν αφεμάσεται με αυτόν τον τρόπο και ε, το, είναι 244 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Εδώ βλέπετε την άδεια που είχε δοθεί αρχικά και που όπως ανέφερα έχει λήξει. Ε, έχουν όμως ξαναρχίσει ε, ανασκαφές εκεί. Αυτή είναι η ζώνη ε, συμβολής προς την πηγή. Αυτή είναι από την υδρογεολογική μελέτη. Βλέπετε την περιοχή με κόκκινο και το νερό το οποίο περνά από πάνω και από κάτω και το οποίο περνά σχεδόν αποκλειστικά στην ε, περιοχή της επιχείρησης, του λατομείου δηλαδή. Ε, δύσκολο να το πιστέψουμε, αλλά τη σήμερα ημέρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης ε, και είναι παράξενο που τόσα χρόνια άντεξε το νερό στη μόλυνση. Τώρα ε, ήδη έχουν γίνει κινήσεις σε βάρος μας ώστε να σιωπήσουμε παρά τις σοβαρές προσφυγές και επιχειρήματά μας. Ε, το 2002 ε, είχε βγει απόφαση ότι η λατόμηση γίνεται χωρίς άδεια. Το 2004 ε, ψηφίσαμε νομοθεσία στην Ιρλανδία για να ρυθμίσουμε το θέμα των λατομείων. Έπρεπε να καταγραφούν, να καταχωρηθούν. Εμείς ε, ζητήσαμε το τοπικό συμβούλιο, το κομιτιακό συμβούλιο να εξετάσει το θέμα το οποίο το 2007 έδωσε ε, μία άδεια στην εταιρεία Woods με 59 όρους. Έδιναν δηλαδή την άδεια με τροποποιήσεις, όρους, προϋποθέσεις πάνω σε ένα ε, πλάνο όμως του 1974 το οποίο κάλυπτε μόνο 5 εκτάρια και το ε, οποίο δεν ισχύει πια. Ε, παραβιάζεται λοιπόν όχι μόνο το Ιρλανδικό αλλά και το κοινοτικό δίκαιο και για, ε, η, περιοχή όπως σας είπα είναι πάνω από 40 εκτάρια. Θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της προφύλαξης που είναι ο ακρογωνίος λίθος της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και ποτέ δεν έγινε ε, ΕΠΕ. Η εταιρεία της Λατόμησης έκανε προσφυγή ε, η κοινότητά μας επίσης ε, ε, κατέθεσε ε, τα επιχειρήματά της και η πρόταση που έγινε είναι η τοπική αρχή να ζητήσει από την εταιρεία του Λατομείου να ζητήσει άδεια ε, για ολόκληρη την περιοχή συνοδευόμενη από μελέτη επίπτωσης περιβαλλοντικού αντίκτυπου. δεν ακολουθήθηκε η συμβουλή αυτή Επίσης από τις 59 προϋποθέσεις ε, έμειναν πολύ λίγες και στο τέλος ε, σχεδόν δεν ε, τροποποιήθηκε τίποτα επί τα βελτίο. Προμηθεύει την τοπική αρχή το λατομείο αυτό. Μπορεί λοιπόν αυτό να παίζει ένα ρόλο εις ό,τι αφορά το αποτέλεσμα σε παραβίαση ε, προς την νομοθεσία ε, μελέτη αντίκτυπου περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ε, σε μια ευαίσθητη περιοχή με τόσο πολλά περιβαλλοντικά θέματα και σε μια περιοχή 40 εκταρίων. Έτσι λοιπόν, εμείς πιστεύουμε στο Watergrass Hill, στην Community Association, ότι δύο κοινοτικέ οδηγίες παραδιάστηκαν, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και εκείνη ε, για την μελέτη περιβαλλοντικού αντίκτυπου. 7.000 ευρώ ε, πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια δαπανήθηκαν για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι ε, οι τοπικές αρχές, η τοπική κοινότητα είναι εκείνη που θα έπρεπε να φροντίσει για το θέμα αυτό της διατήρησης της ποιότητας των υδάτων και στο μέλλον. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή να μας ε, υποστηρίξει στο αίτημά μας να εξεταστεί το θέμα αυτό και να διασωθεί η ποιότητα των υδάτων και το μέλλον. Α, με συγχωρείτε, θέλω να παρουσιάσω και ε, να παρουσιάσω, εάν μπορώ, και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία ε, έχω προσκομίσει. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως μας εξήγησε ο αναφέρον, είναι το θέμα μας η μελλοντική ποιότητα του ποσίμου ύδατος από τη λατόμηση αυτή που λαμβάνει η χώρα. Ευτυχώς δεν έχει μολυνθεί μέχρι τώρα το πόσιμο ύδωρο. Ε, περνώ στις ε, δύο ε, οδηγίες, εκείνη για την οδηγία, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την ε, οδηγία για την μελέτη περιβαλλοντικού αντίκτυπου και αφήνω αυτή για τα οικοσυστήματα, για το πόσιμο ύδωρο και τα πτηνά. Ε, ένα σχόλιο επίσης προς την Επιτροπή. Η ε, εκτίμησή μας για τις οδηγίες αυτές, τις τρεις τελευταίες, κατέληξε ότι δεν υπάρχει παραβίαση, άρα δεν υπάρχει νομική βάση για παρέμβαση της Κομισιόν. Τώρα, εις ό,τι αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και έγιναν διμερείς επαφές μεταξύ αναφερόντων και Κομισιόν, η Κομισιόν τους ενεθάρρυνε να ακολουθήσουν διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την ε, ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα που είναι υποχρεωτική για τις αρχές, όχι για τους ε, πολίτες και να δει τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να αναστραφεί το πρόβλημα ή να μην επεκταθεί το λατομείο περισσότερο και οι αναφέροντες αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία και υπέβαλαν σχετικά έγγραφα στις Ιρλανδικές αρχές. Η Κομισιόν δεν γνωρίζει ακόμα το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας γιατί τα προγράμματα πλάνα στα πλαίσια της οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα πρέπει να, να κοινοποιηθούν μέχρι 22 Μαρτίου 2010 στην Κομισιόν, ε, ένα μήνα δηλαδή, σε ένα μήνα ακριβώς και θα δούμε τότε αν τα μέτρα, μέτρα προφύλαξης, μέτρα διορθωτικά έχουν ληφθεί για τη συγκεκριμένη παροχή του ύδατος στην περιοχή ε, αν δηλαδή έχουν ενσωματωθεί. Ε, τώρα, για την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου επιπτώσεων, το, το κέριο ζήτημα είναι το μέγεθος του λατομείου. Δείχνουν οι διαφάνειές σας αφενός μια περιοχή πυρήνα κεντρική ε, ανασκαφών, λατόμησης δηλαδή, και προφανώς έχουμε μια περιοχή εργασιών που έχει αντίκτυπο σε ευρύτερη περιοχή που δεν καλύπτεται από την άδεια του 1974. Το κέριο ερώτημα είναι αν οι λειτουργίες συνολικά ξεπερνούν τα 25 εκτάρια. Γιατί αν είναι, περιορίζεται σε περιοχή κάτω από 25 εκτάρια, τότε λαμβάνεται απόφαση κατά περίπτωση και κρίνεται αν υπάρχει επίπτωση στο περιβάλλον ή όχι. Αν είναι πέρα από 25 και αν δούμε και τις μελλοντικέ επεκτάσεις, γιατί αυτό είναι το κέριο μέλημα και ανησυχία των αναφερόντων, τότε ξεπερνάει, ε, υπερβαίνεται πολύ το κατόφλι. Τώρα, ε, η Κομισιόν έκανε το συγκεκριμένο ερώτημα στις Ιρλανδικές Αρχές. Ε, σε μια συνάντηση στα μέσα του περασμένου χρόνου και μας είπαν ότι η άδεια έχει εκδοθεί μόνο για 5 εκτάρια πράγμα που συνάδει με αυτό που μας είπε πριν από λίγο και ο αναφέρον. Το ε, βασικό ερώτημα τότε είναι ποιο είναι το καθεστώς. Το, η άδεια μπορεί να είναι ένα κομμάτι χαρτί. Η εταιρεία ε, πληρεί τις προδιαγραφές ε, της άδειας, δηλαδή κάνει λατόμηση μέσα σε αυτή την περιοχή που προβλέπεται στην άδεια. Οι Ιρλανδικές αρχές όχι μόνο το 1974 αλλά και αργότερα ε, είπαν πολύ σαφώς ότι ε, βάσει του Ιρλανδικού δικαίου κάθε λατόμηση ε, κάτω από 5 εκτάρια πέρα από, με πάνω από 5 εκτάρια θα πρέπει να υπόκειται σε μελέτη επίπτωσης περιβαλλοντικών, περιβαλλοντικής. Υπήρξε μια καθυστέρηση από τις Ιρλανδικές αρχές στην απάντηση σχετικά με το μέγεθος του λατομείου. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, αλλά είστε βέβαιοι ότι η Κομισιόν θα επιδιώξει να λάβει τις πληροφορίες που ζήτησε και θα προβεί στη λήψη των αντίστοιχων μέτρων προς τις Ιρλανδικές αρχές. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ που συζητήσατε την αναφορά σήμερα. Είναι πολύ παρήγορο για πολύ κόσμο το γεγονός ότι μπορούν να έχουν προσφυγεί στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Αναφορών και να παρουσιάσουν τα προβλήματά τους ε, όταν δεν ε, εισακούονται στη χώρα τους. Και ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Μπάρι που εκπροσωπεί την Watergrass Community Association για την επιμονή του, το θάρρος του και την τεράστια δουλειά που έκανε για να προετοιμάσει την υπόθεση αυτή. Ε, πραγματικά ε, μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Ε, είδατε και τις διαφάνειες που νομίζω είναι αρκετά πιστικές και εμείς που μένουμε σε αυτήν την περιοχή ανησυχούμε πάρα πολύ για την ποιότητα των υδάτων και αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Όχι μόνο ότι επηρεάζονται οι 800 κάτοικοι του Watergrass Hill, αλλά είναι 50.000 οι κάτοικοι που εφοδιάζονται από αυτή την πηγή υδάτων από αυτό τον υδροφόρο. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν, το πρόβλημα των 50.000 ανθρώπων, αλλά και των δικαιωμάτων τους που παραβιάζονται. Βεβαίως ε, ε, η εταιρεία John A. Woods έχει πολλά λατομεία, όχι μόνο αυτό στην Αγγλία, ε, που ε, λειτουργούν καλά, αλλά στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι θα πρέπει ε, να κοιτάξουμε πρώτα την υγεία των ανθρώπων. Έχοντας ακούσει την Κομισιόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό και ο Μπάρι με διαβεβαιώνει να βεβαιωθούμε για το μέγεθος του λατομείου που είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 5 εκτάρια και μάλιστα υπερβαίνουν κατά πολύ και τα 25, είναι 40 εκτάρια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε παραβίαση των κανονισμών και γι' αυτό θεωρούμε ότι η Water Hill Community Association έχει ένα ισχυρό επιχείρημα στα χέρια της ε, και νομικά αλλά και υγειονομικά. Ε, θα πρέπει να εξαντληθεί το θέμα, να γίνει μια σωστή εκτίμηση των δεδομένων και τέλος να δούμε αν η επιχείρηση αυτή, η J.A. Woods, ε, πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται μόνο να κρίνουμε ε, το γεγονός ότι προσφέρει απασχόληση σε κόσμο. Εδώ έχουμε ένα θέμα υγείας και από ό,τι φαίνεται έχουν λόγο να ανησυχούν. Ευχαριστώ την Κομισιόν, ελπίζω να ε, δοθεί ικανοποιητική απάντηση και πάλι συγχαίρω τον Μπάρι για το θάρρος και την ε, πρωτοβουλία που πήρε ε, και το έργο του στα πλαίσια αυτής της κοινοτικής εταιρείας. Ε, τον Higgins, παρακαλώ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κέρτιν και την ομάδα από το Watergrass Hill για την παρουσίαση που προετοίμασαν. Η εξαιρετική παρουσίαση υπογραμμίζει και πάλι τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι τοπικές κοινότητες που προστατεύουν το περιβάλλον. Ε, κατεξοχήν είναι αυτές και αυτές τα δικαιώματα, δικαιώματα προστατεύουν πάνω από κάθε άλλα. Γιατί όταν μιλάμε για μόλυνση, μιλάμε για κάτι ουσιαστικό ε, που άπτεται της ε, ε, ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος, της υγείας της κοινότητας ε, και της παράδοσης στα παιδιά της κοινότητας, στη νέα γενιά, ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς μόλυνση. Αυτά είναι διαφορετικά θέματα από τα εμπορικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης, η κυβέρνηση, το κράτος πολλές φορές ε, είναι εμπλεκόμενη με σύγκρουση συμφερόντων ε, προς ε, τα συμφέροντα αναπτυξιακών εταιριών κλπ ή κατασκευαστικών εταιριών. Ε, νομίζω ότι δεν κατάλαβα 100% αυτά που μας είπε η Κομισιόν. Θα διαβάσω όμως την τεκμηρίωση σχετικά για να ενημερωθώ. Σίγουρα όμως η περιοχή αυτή είτε είναι 5 εκτάρια είτε παραπάνω δεν είναι το κέριο ζήτημα. Η κρίσιμη περιοχή είναι το μέγεθος της περιοχής που παγιδεύεται γιατί αν η λειτουργία μιας επιχείρησης περιορίζεται σε δύο εκτάρια αλλά διαταράσει το περιβάλλον ή το μολύνει, εν προκειμένου ε, τα ύδατα, επηρεάζει μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης ότι μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη απειλούμενη περιοχή. Πρέπει να κατησχύσει η κοινή λογική εδώ. Όταν ε, υποβάλλεται μια υπόθεση με τεκμηρίωση με τόσο σαφή τρόπο όπως σήμερα, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Τα στοιχεία επιτόπου μιλούν από, το, από μόνα τους. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι είναι ο θεματοφύλακας ε, του περιβάλλοντος και προστάτης των βέλτιστων πρακτικών πέρα από τοπικά συμφέροντα, ε, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να προστατέψει σε αυτή την περίπτωση την τοπική κοινότητα. Ευχαριστώ. Ε, is there anybody, ε, υπάρχει κανείς που θα ήθελε να μιλήσει. Ε, προτείνουμε τότε να γράψουμε, να, να κάνουμε μια επιστολή προς την προς το Ιρλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος ε, περιμένοντας ε, κάποια σαφή απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα. Μιας και έχουμε σαφή παραβίαση ό,τι αφορά τα 25 εκτάρια, τα 5 εκτάρια που υπερβαίνουν τον επιτετρό αριθμό. Ε, προχωρούμε λοιπόν στην επόμενη που προέρχεται από τη Γαλλία και αφορά την κατασκευή γέφυρας πάνω από το Λίγυρα ανατολικά από την Ορλάνη.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 Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το ενδιαφέρον που δείξατε για την αναφορά μας, η οποία αντιτίθεται σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας γέφυρας και περιφερειακής οδού γύρω από την Ολεάνη. Αυτό αποφασίστηκε το 2007 στα πλαίσια ενός σχεδίου χωρικής συνοχής που αφορούσε την περιοχή ανατολικά της Ορλεάνης και συγκεκριμένα την κατασκευή γέφυρας πάνω από το Λίγυρα εκεί. Εμείς αντιτιθέμεθα σε αυτό το σχέδιο γιατί θεωρούμε ότι το σχέδιο βασικό κύριων προσανατολισμών δεν είναι αρκετά σαφές και επίσης δεν ελήφθησαν υπόψη οι δυνατότητες ή εναλλακτικές. Καταρχάς, όσον αφορά το σχέδιο χωρικής συνοχής ΣΚΟΤ, θα ήθελα να πω ότι δεν ληφθήσαν υπόψη θέματα όπως ε, η αντιμετώπιση της μόλυνσης, ε, του θορύβου, της προστασίας του τοπίου κλπ. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας γέφυρας η οποία είναι αντίθετη σε όλες τις αρχές μας. Πρόκειται για μια ευαίσθητη περιοχή και η γέφυρα θα περνά από χώρες, από περιοχές με που έχουν προστατευτεί στα πλαίσια του προγράμματος Natura 2000. Και θα δημιουργηθεί μόλυνση τόσο περιβαλλοντική όσο και ηχητική αυτό που βλέπουμε είναι ότι η γέφυρα αυτή θα είναι για μια γέφυρα παράκαμψης η οποία θα επιτρέπει την διέλευση των βαρέων οχημάτων που κινούνται από τη Γαλλία προς τη Βαρκελόνη στον Νότο. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό τεχνικά. Επίσης, υπενθυμίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία όσον αφορά την Ορλεάνη, η οποία δεν ελήφθη υπόψη, όπως επίσης δεν ελήφθη υπόψη και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ειδικά όσον αφορά την προστασία της περιοχής αυτής, η οποία προστατεύεται μεταξύ άλλων και από τις οδηγίες Habitat, τις οδηγίες για τα πτηνά, αλλά και πρόκειται και για τόπο πολιτισμικής κτηνονομιάς που προστατεύεται από τη Σύμβαση UNESCO. Η οργάνωσή μας θα ήθελε να τονίσει την κατάσταση και επίσης να τονίσουμε ότι δεν έχει γίνει μελέτη επιπτώσεων περιβαλλοντικών και άλλων. Οπότε, εμείς θεωρούμε ότι αν στόχος μας είναι η διατήρηση της ε, δικαιοφικιλότητας, τότε δεν μπορεί να γίνει αυτό το, αυτή η γέφυρα η οποία θα είναι θα αντιτίθεται στην νομοθεσία που ήδη ισχύει. Ειδικά τους στόχους 4, 5 που αφορά τις μεταφορές, 7 βιοπικιλότητα, Επίσης να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν σεβάστηκε ούτε τον περιφερειακό χάρτη που ισχύει για την περιοχή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπήκαν οι περιοχές αυτές σε και κομπλέ στο ΣΚΟΤ, το σχέδιο χωρικής συνοχής, χωρίς καμία διαβούλευση ή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται η τοπική αυτοδιοίκηση της Ορλεάνης προσπαθεί να κλείσει όλη την κυκλοφορία μέσω Ορλεάνης από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή σκέφτονται να καταργήσουν ορισμένες διαβάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν την μεγαλύτερη κίνηση. Επίσης αρνούνται να επεκτείνουν την ε, γραμμή προς το ΣΕΣΥ προκειμένου να βοηθηθεί η κατάσταση καθώς επίσης και τη βελτίωση των σιδηροδρομικών γραμμών. Και εμείς από την πλευρά μας είπαμε ότι θα έπρεπε να μην γίνει αυτή η γέφυρα. Στη διαβούλευση που είχε γίνει για το ΣΚΟΤΕ είχε αναφερθεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνει διάβαση του ΣΕΣΥ. αλλά τελικά αποφασίστηκε η δημιουργία της γέφυρας, γι' αυτό το λόγο η οργάνωσή μας έκανε πρόσφυγη. Παρόλα αυτά όμως εγκρίθηκε τελικά το ΣΚΟΤ τον Δεκέμβριο του 2008. το αίτημά μας παραμένει το ίδιο. Ζητάμε αυστηρό σεβασμό των περιβαλλοντικών κανόνων, ειδικά των στόχων 4, 5, 7 του περιβαλλοντικού συμφώνου του Προεδρικού στη Γαλλία και την απόσυρση του σχεδίου δημιουργίας γέφυρας ανατολικά της Ορλεάνης, όπως προβλέπεται από το σχέδιο χωρικής συνοχής ΣΚΟΤ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από την Κομισιόν, ο κύριος Βάντερ ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κάποιες εξηγήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο φάκελο Ήδη έγινε παρουσίαση, οπότε να κάνω μια σύνοψη. Η προσφυγή αφορά τη δημιουργία μιας γέφυρας πάνω από το Σεσί Κομπλέ στο Λίγυρα. Θεωρούν ότι δεν είναι αποδεκτή μια τέτοια κατασκευή ειδικά εφόσον η περιοχή του Λίγυρα καλύπτεται από την προστασία των, οδηγών, των οδηγιών Habitat και οδηγία για τα πτηνά, καθώς επίσης και από την UNESCO. Πρόκειται για σχέδιο που αφορά την απεμπλοκή των πόλεων, των αστικών κέντρων. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε ως ανάλυση. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα σχέδιο χωρικής ε, συνοχής ΣΚΟΤ, το οποίο εγκρίθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση στις 18 Δεκεμβρίου του 2008 και όπου συμπεριλαμβάνονται οι γενικοί προσανατολισμοί για τα επόμενα 20 έτη. Βεβαίως χρειάζονται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατασκευή της γέφυρας. Άρα η κατασκευή της γέφυρας παραμένει καθαρά σε υποθετικό πλαίσιο. Και πρόσφατα τον Νοέμβριο μας επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει γίνει καμία άλλη ενέργεια και δεν πρόκειται να γίνει κάτι πριν το 2020. Τώρα, αν κάποια στιγμή ληφθεί απόφαση για κατασκευή της γέφυρας θα έπρεπε να γίνει εκτίμηση επιπτώσεων που θα αφορά και τις οδηγίες Habitat και οδηγία για τα πτηνά και τότε θα έπρεπε να γίνει και δημόσια διαβούλευση. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. εν συντομία κάποιες σκέψεις. Το νέο στοιχείο είναι ένα διοικητικό έγγραφο που προχωρά στο θέμα της σκοπιμότητας της γέφυρας και πρόκειται για το έγγραφο της 18ης Δεκεμβρίου του 2008. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το θέμα της ε, παράκαμψης της Ολεάνης ε, δεν είναι νέο. Ήδη είχαμε μία αναφορά από το 2004 που είχε συζητηθεί το 2005 από την Επιτροπή. Άρα με το θέμα ασχολούμαστε εδώ και πάνω από έξι χρόνια χωρίς να έχουμε καμία εγγύηση όσον αφορά τους κινδύνους που παραμένουν για τη βιοπικιλότητα. Μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για υποθετικό σχέδιο, όμως θα είναι κάτι που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη βιοπικιλότητα και το περιβάλλον. Εδώ και έξι χρόνια λοιπόν αυτό το σχέδιο παραμένει υποθετικό αλλά πιθανό μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Θα έπρεπε, μετά από έπρεπε, θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει με το σχέδιο αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι το 2009 είχαμε λάβει και δεύτερη αναφορά επί του θέματος Οπότε εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε προχωρήσει όπως θα έπρεπε και ότι οι γαλλικές αρχές επιμένουν στο ότι ο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το έργο και παραμένει υποθετικό και μιλάνε για ορίζοντα 2020 αλλά δεν κάνουν τίποτα πέραν αυτού. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε η Επιτροπή μας να στείλει μια επιστολή στις γαλλικές αρχές και στις αρμόδιες αρχές ειδικά στις αρχές που εκπώνησαν το σχέδιο χωρικής συνοχής, το ΣΚΟΤ, προκειμένου να υποχωρήσουν σε αυτό το σχέδιο που αφορά προστατευόμενες γεωγραφικές ζώνες. Και σας υπενθυμίζω ότι η προστασία της βιοπικιλότητας όπως αναφέρεται στην οδηγία Habitat δεν αφορά μόνο τα projects, τα προγράμματα αλλά και τα σχέδια. Άρα και το σχέδιο χωρικής συνοχής πρέπει επίσης να σέβεται και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας Habitat. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ούκεν, το λόγο. Uh, sorry, sorry. Η <laughs> ε, κυρία Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που ήρθαν μέχρι εδώ για να μας εξηγήσουν την αναφορά τους. Όντως πρόκειται για δύσκολο θέμα γιατί παραμένει σε επίπεδο σχεδίου. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε επίσης εδώ το γαλλικό κράτος και την επιτροπή μας εδώ η οποία μπορεί να κάνει μόνο συστάσεις. Μέχρι σήμερα το σχέδιο αυτό δεν έχει προχωρήσει. Παραμένει, όπως υπόθηκε και από την κυρία Μπελιέ, σε καθαρά υποθετικό πλαίσιο. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να περνάμε χρόνια συζητώντας το θέμα. Καταλαβαίνω επίσης τα επιχειρήματα της κυρία Μπέλιε για το περιβάλλον. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σχέδιο και τίποτα παραπάνω. Καταλαβαίνω τους αναφέροντες που τους ενδιαφέρει προσωπικά το θέμα και μας λένε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προσέξουμε τι αναφέρουν οι οδηγίες Habitat και οδηγίες για τα πρινά. Και συμφωνώ. Αλλά από τη μία πλευρά κάθε φορά παραπονιόμαστε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξα τα κράτη-μέλη και από την άλλη όποτε προτείνουν κάποια σχέδιο αμέσως αντιτιθέμεθα. Βεβαίως πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις και αναλύσεις αντικτύπων. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν λέω λοιπόν εγώ ότι είμαι κατά, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα πρέπει να περιμένουμε την ανάλυση αντικτύπου. Και τότε θα μπορούμε να λάβουμε θέση και εμείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την εργασία που έγινε για το θέμα αυτό και πρέπει να σας πω ότι εγώ ε, συμμετείχα σε μια αποστολή fact-finding πριν από δυόμιση χρόνια και ε, πήγαμε στην Ορλεάν ε, και στην περιοχή αυτή του Λίγυρα. Και όσον αφορά την ομάδα μου θα ήθελα να σας πω ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ε, ότι αυτά τα, τα έργα ε, πραγματικά ε, μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη ότι δηλαδή δημιουργούν ε, θέσεις απασχόλησης χωρίς να μας απασχολεί καθόλου το θέμα της πράσινης ανάπτυξης, πράσινης ε, δράσης. Εγώ πρέπει να σας πω, όταν πήγα εκεί, με εξέπληξε ιδιαίτερα το γεγονός, γιατί η περιοχή είναι θαυμάσια, είναι εξαιρετική. Ε, εκεί Πώς να σα το πω, ε, πραγματικά ε, όταν έχουμε μια τόσο ε, όμορφη περιοχή είναι ανεξήγητα όλα αυτά. Σκεφτήκαμε, μα τι γίνεται με όλη αυτή την κυκλοφορία, πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν τόσο πολλά οχήματα. Και όσον αφορά τις υποδομές, ε, ε, ε, και το τι. Τώρα, εκεί είδαμε τι δυνατότητε υπάρχουν για τη χρησιμοποίηση των υποδομών. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω τι γίνεται με τι ανάγκε. Αυτό είναι θέμα των τοπικών αρχών. Το μόνο που θέλω να σα πω είναι ότι αισθάνομαι έκπληξη για το γεγονό ότι μιλάμε για τέτοια κλίμακα έργα σε τέτοιε περιοχέ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για άλλε ζώνε. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να γίνονται μελέτε, οι οποίε βεβαίω είναι απαραίτητε και να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σεβαστοί οι κανόνες και οι προϋποθέσεις της οδηγίας Natura. Η ανάλυση λοιπόν των συνεπειών, ο αντίκτυπος των, ε, η μελέτη αντικτύπου θα πρέπει να είναι συνολική, να εξετάζεται συνολικά ο αντίκτυπος. Άρα θα θέλαμε να μάθουμε τον αντίκτυπο σε όλη την περιοχή του Λίγυρα και όχι μόνο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο έργο, αν θέλετε, και σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, αλλά στο σύνολό του. Δηλαδή, Εάν εγώ ήμουν από την περιοχή αυτή, ειλικρινά θα αγωνιζόμουν με νύχια και με δόντια για να υπερασπιστώ ε, το δικαίωμα να έχουμε μια τέτοια περιοχή η οποία είναι πόλος, πόλος έλξης τουριστών που χαρακτηρίζεται από φυσικές ομορφιές, ε, από το περιβάλλον. Ε, θα, θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εγώ διαφωνώ με το να τσιμπεντοποιούμε τα πάντα ε, τώρα βέβαια δεν είμαι εγώ αυτή που ε, πρέπει να τοποθετηθώ επί της ουσίας. Απλά και μόνο ήθελα να σε εκφράσω ορισμένες σκέψεις μου και κυρίως την έκπληξή μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όκεν. Ε, υπάρχει μια πρόταση από την κυρία Πελιέ, από την κυρία Μπελιέ να στείλουμε ένα έγγραφο στις γαλλικές αρχές, στην περιοχή, στην, στις τοπικές αρχές. τι θα πρέπει, καταρχήν συμφωνούμε όλοι, όχι, αυτό πρέπει να αποφασιστεί ε, ε, τέθηκε μία πρόταση. There was a suggestion by Mrs. Bellier concerning the... Ε, Υπήρξε μία πρόταση της κυρίας Μπελιέ για αποστολή επιστολής προς τις αρχές της Νέας Ορλεάνης. προκειμένου να λάβουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό το πρόγραμμα. Θέλετε να σταλεί αυτή η επιστολή ή όχι. Είναι κάτι επί το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα να στείλουμε επιστολή, αλλά τι θα μπει μέσα. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνει ανάλυση αντικτύπου. Αλλά άμα πρόκειται να στείλουμε επιστολή, τι θα γράψουμε. Και να πω στην κυρία Μπελιέ ότι όλη η Γαλλία είναι πανέμορφη. Στην κυρία Άουκεν, μας συγχωρείτε. Europe is beautiful, I must say. <laughs> Uh, uh, anyway, Αυτό που προτείνω είναι να υπενθυμίσουμε στις αρμόδιες αρχές με την επιστολή αυτή τις υποχρεώσεις τους από την οδηγία Habitat όσον αφορά την προστασία των φυσικών βιοτόπων και της βιοπικιλότητας και την ε, συμβατότητα αυτού του σχεδίου με τις ε, διατάξεις ε, της οδηγίας και αν υπάρξει ανάλυση αντικτύπου θα έπρεπε να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει ισορροπία και συμβατότητα των όσων προβλέπονται από το ΣΚΟΤ με τις διατάξεις ε, των οδηγιών. Μια ερώτηση. Αν ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση του θέματος σαν να έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή, μήπως τελικά το κάνουμε πιο υπαρκτό πώς να το θέσω αλλιώς. Του δίνουμε υπόσταση. Προτείνω την εξή προσέγγιση. Η οδηγία Habitat αναφέρει ότι οι στόχοι προστασίας της ποικιλάτητας αφορούν τα σχέδια και τα έργα, plans and projects. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι δεν έχει εγκριθεί το έργο και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη μελέτες. Εμείς προτείνουμε να μην αναφερθούμε στο έργο, το project, αλλά στο σχέδιο το οποίο εγκρίνθηκε τέλη του 2008, πρόσφατα δηλαδή και αφορά τον αστικό σχεδιασμό και προβλέπει την πιθανότητα κατασκευής αυτής της γέφυρας. Οι αρμόδιες αρχές λοιπόν θα λάβουν υπόψη αυτό το σχέδιο προκειμένου να κάνουν τις μελλοντικές τους, ε, τα μελλοντικά τους βήματα όσον αφορά τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να αναφερθούμε. Ε, ε ευχαριστώ πολύ. Ε, it's up to us Uh, this Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να στείλουμε μια ευγενική επιστολή που να ζητά διευκρινήσεις. Διαφωνείτε από αυτού. Νομίζω ότι αυτό θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές και θα είμαστε και ευγενικοί προς τις αρχές γιατί πρόκειται περί σχεδίου απλώς που μπορεί ποτέ να μην πραγματοποιηθεί. Ωραία. Oh. Θέμα 16. Θέμα 16. Ολιβιέρ Περόν, ε, ο αναφέρον. Σε σχέση με μια πολεοδομική άδεια για αναπτυξιακό έργο. Ο Ολιβιέ Περόν δεν είναι εδώ. Να προσπαθήσετε λοιπόν να μα εξηγήσετε, ο κύριος Παντεστέγγε θα μα εξηγήσει. Κύριε Πρόεδρε, να σας συνοψίσω την κατάσταση. Ο αναφέρον ε, ε, αναφέρεται στην έκδοση πολυδομικής άδειας για την κατασκευή 23 συλλογικών κατοικιών, 30 μεμονωμένων κατοικιών και ενός οικού ευγυρίας. Ε, σε μια περιοχή που βρίσκεται εντό μια προτευόμενη περιοχή για τα πτηνά, στα πλαίσια τη ε, ε, οδηγία για τα πτηνά. Ο αναφέρον αναφέρεται στι αρνητικέ επιπτώσει επί των αρλικών και σε παραβίαση τη οδηγία για τα οικοσυστήματα. Υπήρξε λοιπόν προσφυγή κατά της έκδοσης πολεοδομικής αδείας ενώπιν του Διοικητικού Δικαστηρίου της Νάντης ε, αλλά ε, επειδή ε, η περιοχή αυτή ορίστηκε ως προστατευόμενη ζώνη μετά την έκδοση της άδεια, στη συνέχεια έκανε, έκανε ξέφεση κατά της απόφασης αυτής κτλ. Λοιπόν, να σας πω, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της οδηγίας για τα πτηνά, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγουν στις δικές προστατευόμενες ζώνες τη ρήπανση ή την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, καθώς επίσης και τις τις ε, ε, ενοχλήσεις που μπορεί να προκληθούν στα πτηνά. Σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι ζώνες ειδικής προστασίας, οι οποίες δεν είχαν οριστεί ως τέτοιες, αλλά που θα έπρεπε να έχουν οριστεί, θα πρέπει να ωφελούνται από το ίδιο καθεστώς προστασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η, επέκταση τη ε, προστατευόμενη ζώνη, συμπεριλαμβάνοντα και την περιοχή αυτή, είχε υποβληθεί στο, στο τοπικό συμβούλιο πριν εκδοθεί άδεια, τρει μήνε. Οι ε, ενδιαφερόμενοι ε, κλάδοι όμω για την... Οι ε, μάλλον τομείς από την, από τη συγκεκριμένη κατασκευή του έργου συμπεριλαμβάνονται στην προστατευόμενη ζώνη. Και επομένως εφαρμόζεται σαφώ και ισχύει η οδηγία για τα πτηνά. Να σα μιλήσω τώρα για τις τελευταίε εξέργου αυτό από την τελευταία προφορική ανακοίνωση στην Επιτροπή Αναφορών στι 21 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ενημερωτική επιστολή στι γαλλικέ αρχέ, ζητώντα ε, να περιγράψουν διεξοδικά την κατάσταση, τόσο όσον αφορά το ίδιο το έργο, αλλά και τι δικαστικέ και διοικητικέ επιτυχίε. Εξάλλου, ο φάκελος ε, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της ε, ε, τελευταίας συνεδριάσης, συνεδρίασης που έγινε στο Παρίσι και τότε πήραμε καλέ ειδήσει, αν θέλετε, γιατί οι γαλλικές αρχές μας ενημέρωσαν για το ότι ε, το σχέδιο αυτό, το έργο αυτό ε, είχε εγκαταληφθεί, ότι ένα ε, μέρος του τμήματος, το ένα μέρος της περιοχής το είχε εξαγοράσει το, τοπικό συμβούλιο και ένα άλλο μέρος της συγκεκριμένη περιοχής θα μπορούσε να αγοραστεί από μία άλλη κοινότητα έτσι ώστε να γίνει ένας, ένα πάρκο. Ζητήθηκε η γραπτή επιβεβαίωση όλων αυτών των πληροφοριών και θα σας τηρήσουμε ενήμερους. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, θα ήθελε κάποιος να μιλήσει. Ε, ε, Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κλείσει η αναφορά προ στιγμή, εφόσον δηλαδή δεν έχουμε πάρει ακόμα ε, τα συγκεκριμένα αυτά έγγραφα, αλλά νομίζω ότι μάλλον θετικέ οι εξελίξει και στην ουσία ε, συμφωνούν και με τι δικέ μα συνομιλίε με του αναφέροντε όταν ήρθαν ε, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Νομίζω λοιπόν ότι μάλλον καλέ είναι αυτέ οι ειδήσει και σα ευχαριστούμε. Ε, κύριε Κύριε Πρόεδρε, και εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, τουλάχιστον μέχρι να πάρουμε γραπτές και επίσημες πληροφορίες από το Δημαρχείο και από την τοπική, από αυτοδιοίκηση. Με τη γραπτή απάντηση μπορούμε να αποφασίσουμε είτε να δηλώσουμε ότι, ότι θα κλείσουμε την αναφορά είτε να συνεχίσουμε. Ωραία. Συμφωνώ με την άποψη των συναδέλφων. Και ε, θα πάρουμε πληροφορίες από του αναφέροντες που ζήτησαν συγγνώμη για το γνώστο. ότι δεν παρευρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά ήταν πολύ... δεν είχαν χρόνο, ήταν πολύ σύντομε σύντομο το χρονικό διάστημα. Μα ζήτησαν λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι να έχουμε και γραπτή επιβεβαίωση. Νομίζω ότι πράγματι ε, είναι λογικό να περιμένουμε λίγε εβδομάδε. Και αν χρειαστεί, σε μια προσεχή συνεδρίαση, αν δεν πάρουμε γραπτή επιβεβαίωση, ίσω θα μπορούσαμε έτσι να. Βεβαίω, ε, στην ε, στην ικανοποίησή μα για τι εξελίξει, αλλά ε, να, να σπρώξουμε κάπω την όλη υπόθεση, να πάρουμε γραπτή επιβεβαίωση και ταυτόχρονα να σας πω, μεταφέρω την άποψη των αναφερόντων και ήθελα να σας πω ότι τόνισαν το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών στο ζήτημα αυτό, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν αμεληταίος ε, ε, και σίγουρα έχει σχέση με αυτή την ευτυχή έκβαση που όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εδώ βρισκόμαστε απόλυτα σε μια περίπτωση όπου ανθρώπινες δραστηριότητες, οικονομικές δραστηριότητες και ποιότητα της φύσης και τα τρία αυτά στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και αλληλεξαρτώμενα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ότι είμαστε σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε περιμένοντας ακόμη πιο θετικές ε, ε, ε εκδηλώσεις από τη μεριά των αναφερόντων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την επόμενη, αριθμός 17. Ε, πρόκειται για αναφορά του κυρίου Νίλσεν με στόχο ένα συγκρότημα εξοχικών κατοικιών στη Δανία που πιστεύετε ότι παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Ε, είναι εδώ από την μεριά της Επιτροπής ε, η κυρία Πλάνκ. Παρακαλώ. Η κυρία Πλάνκ. Thank you, Madam σας ευχαριστώ. Από μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπήρξε διαμαρτυρία σε σχέση με το γεγονός ότι οι δανεικές αρχές έχουν επιτρέψει ε, αυτή, την, ε, ε, αυτή, αυτή την οικοδόμηση πρώτα 20 και μετά και άλλων εξοχικών κατοικιών σε αυτό το νησί. Το νησί αυτό είναι, έχει 4 χιλιόμετρα μήκο και 3 χιλιόμετρα πλάτο. και η Επιτροπή μπορεί να σε επιβεβαιώσει ότι ολόκληρο το νησί Άρο έχει οριστεί από τη Δανία ως μέρος του δικτύου Natura 2000. Ο χαρακτηρισμός έγινε ε, με βάση τις δύο οδηγίες, τη μία για τα οικοσυστήματα, οικοτόπους και η άλλη για τα πουλιά. Επίσης είναι θεωρείται υγροβιότοπος ε, εθνικής σημασίας με βάση τη σύμβαση Ραμσάρ. Οπότε πρόκειται για περιοχή, από ό,τι φαίνεται, που ε, προστατευόμενη οικότοποι και ε, πτηνά και υπάρχουν τρία είδη τα οποία είναι τα κυρίως προστατευόμενα μεταξύ του είναι και το σύρκους αερογόνησους το Δανικό Κοινοβούλιο ανοίχθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης με τη συμφωνία τους, πρώτα 20 μετά 12 ε, και μια καινούρια οδηγία προτάθηκε ε, για τα 12 αυτά εξοχικά. Και ο αναφέρον ε, ανησυχεί για αυτές τις άδειες εφόσον θεωρεί ότι τα εξοχικά ε, πηράζουν το περιβάλλον στο μικρό νησί Άρο και θα είναι επιζήμια για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος. 17% το 70% ε, των ε, περιοχών καλύπτονται από την Νατούρα και επειδή δεν ε, προβλέπ... και δεν προβλέπεται, απαγορεύεται δεν απαγορεύεται όμως ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτά τα πλαίσια. Όμως οποιαδήποτε σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται σε μελέτη επίπτωσης περιβαλλοντικής ε, και θα πρέπει να ισχύει και η οδηγία για τους οικοτόπους που προβλέπει ότι προγράμματα που δεν συνδέονται με τη διαχείριση της περιοχής αλλά που είναι πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά την περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει για την διατήρηση της περιοχής. Όλοι γνωρίζουμε την αξία της ε, περιοχής ε, και την προστασία της φύσης. Οι ιδανικές αρχές λοιπόν ε, εκτίμησαν τον πιθανό αντίκτυπο των εξοχικών κατοικιών πάνω σε αυτό το νησί. Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση των 20 εξοχικών, η Κομισιόν εξέτασε την υπόθεση και θα ήθελε να σημειώσει ότι σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες από τις δανεικές αρχές το άρθρο 6 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους ε, έχει τηρηθεί και, στην, ε, και η αξιολόγηση έγινε προβλέποντας όρους ε, για την μετέπειτα διαδικασία σχεδιασμού και οικοδόμησης. Επίσης, η ΕΠΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2001 κάθετο 42 ΕΕ, έχει ε, χρησιμοποιηθεί ε, για την χωροταξική οδηγία. Με βάση τις πληροφορίες που πήρε η Κομισιόν από τις Δανικές Αρχές, δεν σημειώνεται παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, στα πλαίσια της διαδικασίας για την προτινόμενη ανάπτυξη. Και σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση του Αυγούστου του 2008, οι αναφέροντες έδωσαν συμπληρωματικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνοντας μια ένσταση στην πρόταση για μια νέα ε, χορταξική οδηγία για πρόσθετες 12 ε, εξοχικές κατοικίες οι δανεικές αρχές εκλήθησαν να δώσουν ε, συμπληρωματικές πληροφορίες και η Κομισιόν ειδικότερα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων και των σωρευτικών επιπτώσεων από την προσθήκη των 12 εξοχικών κατοικιών. Η Κομισιόν ζήτησε από τις δανεικές αρχές να εξηγήσουν πώς θα διασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις δύο οδηγίες οικοτόπων και πτηνών και πώς θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει σημαντική διατάραξη του περιβάλλοντος ή ζημιά στους οικοτόπους και στα είδη ε, που καλύπτονται ε, στην περιοχή αυτή. Η Κομισιόν ενημερώθηκε ότι δύο ΕΠΕ ε, έλαβαν χώρα. Οι δανεικές αρχές εξήγησαν τα συμπεράσματα από αυτές τις ΕΠΕ, εξήγησαν τις ανησυχίες που εκφράζονται για το συγκεκριμένο νησί που είναι ένα νησί στο οποίο έρχονται πολλοί αλληλείς και φέρνουν τα ζώα τους, σκύλους για παράδειγμα, που τρέχουν πάνω στο νησί και που θα μπορούσαν και εκείνοι να επηρεάσουν την ε, ζωή των πτηνών στο Άρο Κάλφ, ε, που είναι μια σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή των πτηνών. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και ευρήματα, οι δανεικές αρχές πρότειναν κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ε, επόμενο διεξοδικό σχεδιασμό και είναι πολλά μέτρα. Για παράδειγμα, ε, ε, οι περιοχές αυτές που θα είναι οι εξοχικές κατοικίες θα είναι ανοιχτέ αν και θα υπάρχουν φράχτες με θάμνους που θα προστατεύουν. Οι αναπτυξιακές εργασίες θα λάβουν χώρα εκτός της περίοδου αναπαραγωγής μετά τις 15 Ιουλίου πριν από την 1η Μαρτίου. Έτσι λοιπόν οι φράχτες κατά μήκος του δρόμου ε, μεταξύ των χωριών δύο χωριών ε, θα διατηρηθούν, ούτω ώστε να μειωθεί ο θόρυβος που προκύπτει ίσως από την κυκλοφορία στην ε, νοτιοδυτική περιοχή και θα, υπάρξει, θα ξεκινήσει και μια ενημερωτική εκστρατεία με φυλάδια ε, σχετικά με την προστασία της ορνηθοπανίδας στο Άρο και στο Άρο Κάλφ η σήμανση για την απαγόρευση της πρόσβασης κατά τη διάρκεια της περίοδου αναπαραγωγής θα αναθεωρηθεί και θα εξεταστούν τρόποι βελτίωσής της. Ε, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής ενός πιο αποτελεσματικού φράχτη στο φυσικό καταφύγιο Αροκάλφ που θα εμποδίζει την είσοδο σκυλιών και γατών και θα εξεταστεί η ανάγκη για πρόσθετα μέτρα στο γυλιόμενο σχεδιασμό Natura 2000. Ε, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα αυτά, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα έχει ληφθεί η αναγκαία μέρη σχετικά με του οικοτόπου και τα είδη στην νομοθεσία Natura 2000 για τα τις ε, αρχές αυτές. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι σορευτικές επιπτώσεις αυτού του είδους ανάπτυξη σε κάθε μελλοντικό σχεδιασμό για την εν λόγω τοποθεσία και την ανάγκη να υπάρξει διαχείριση των πιέσεων για δραστηριότητες αναψυχής. Οι αρχέ έχουν ενθαρρυνθεί να αναπτύξουν ένα σχέδιο διαχείρισης για τη συγκεκριμένη τοποθεσία ως μέσο συμφιλίωσης των δραστηριοτήτων αναψυχή με τη διατήρηση των ειδών και χαίρομαι μπορώ να σας πω ότι το σχέδιο αυτού του σχεδίου διαχείρισης μαζί με άλλα σχέδια διαχείρισης άλλων περιοχών Ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2010 και θα ε, πρόκειται να γίνουν διαβουλεύσεις με τις ε, δημοτικές αρχές στη Δανία. Ε, αυτά τα σχέδια ε, σχεδίων πλάνων διαχείρισης υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορούμε, μπορεί όποιος ενδιαφερόμενος είναι να τα δει από εκεί. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, βεβαίως, κυρία Χάουκεν. Θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά την Επιτροπή, γιατί νομίζω ότι πραγματικά ήταν αποτελεσματική αυτή η εργασία κατά από πολλέ ε, απόψει. Γιατί εδώ έγιναν μια σειρά από συναντήσει, αν θέλετε, και σε προσωπικό επίπεδο. Μπορώ να σα πω ότι ε, ε, σχηματίσαμε μια ιδέα κατά πόσο θα έπρεπε να γίνουν δηλαδή αυτέ οι εξοχικέ κατοικίε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, εδώ έγινε μία σειρά από ε, συζητήσεις και στην Δανία. Ήταν ιδιαίτερα έντονες θα έλεγα. Πάντως συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα συμπεράσματα ε, ε, τα οποία ακούσαμε εκεί και με βάση όλα αυτά τα στοιχεία. Επομένως δεν έχετε αντίρρηση. You don't have any objections. Okay then. Uh, so, let's hope that... Uh, Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτές οι υποσχέσεις θα εφαρμοστούν και δεν θα γίνουν... Α, γιατί αυτό είναι μια, ένα ενδεχόμενο, να μπορεί να μην γίνουν αυτές οι 12 πρόσθετες εξοχικές κατοικίες στην περιοχή. Ε, concerning ε, road that Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αναφορά που έχει να κάνει με ένα αυτοκινητόδρομο μεταξύ Κίπλεφ και Σόντερμπορκ στη Δανία. Uh, uh, λοιπόν, να ακούσουμε την Επιτροπή, τον κύριο Κάσμαν. Όχι, δεν είναι ο κύριος Κάσμαν. Ζητώ συγγνώμη. Είναι ο συνάδελφός μου, κύριε Πρόεδρε η συνάδελφό μου, η Σίλβια Άιλ, η οποία θα απαντήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται λοιπόν για μία αναφορά που αφορά ένα σχεδιαζόμενο αυτοκινητόδρομο ανάμεσα στο Κίπλεφ και στο Σόντερβολκ στη Δανία. Ο αναφέρον εξέφρασε ανησυχίε όσον αφορά ε, την επίπτωση του σχεδίου σε προστατευόμενε περιοχέ που βρίσκονται κοντά στο σημείο αυτό. Έγινε εκτενή αξιολόγηση από την Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας επί παραβάση. Το σχέδιο αυτό επίσης και το έργο ε, συζητήθηκε σε μια ε, συνεδρίαση με τις δανεικές αρχές. Σαν αποτέλεσμα, οι αρχές της Δανίας συμπλήρωσαν τις αρχικές τους επιπτώσεις και προέβησαν συμπληρωματική αξιολόγηση επιπτώσεων και εισήγαγαν άλλα μέτρα ε, έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο συγκεκριμένα με την οδηγία για τα οικοσυστήματα και τα άγρια πτηνά. Άρα λοιπόν η Επιτροπή έλαβε απόφαση στις 19 Μαρτίου του 2009 να κλείσει την υπόθεση και δεν υπήρξαν συμπληρωματικές πληροφορίες στο μεταξύ που να έφτασαν ε, στην Επιτροπή σε σχέση με το έργο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Όκεν. Κοιτάξτε, εδώ δεν θα είμαι τόσο ευγενική, γιατί το πρόβλημα εδώ έχει να κάνει με το εξή. Δηλαδή, έχουν γίνει μελέτε, υπάρχουν μελέτε που δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Για παράδειγμα, να δούμε τι σορευτικέ επιπτώσει από την αύξηση τη κυκλοφορία. Γιατί μετά από τα ε, έργα αυτά, καταλαβαίνετε, θα υπάρξει τρομερή συγκέντρωση της κυκλοφορίας. Ε, που, που θα, και εδώ μιλάμε για μια ζώνη η οποία ε, είναι προστατευόμενη στα πλαίσια του Natura 2000. Και εμεί έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε την οδηγία. Λοιπόν, για να σεβαστούμε την οδηγία πρέπει να πραγματοποιηθεί μελέτη για τι ορευτικέ επιπτώσει. Δεν το ζήτησε η Επιτροπή, ούτε την έκανε τη μελέτη αυτή η Δανία. Ε, λοιπόν, ένα από τα πιο προφανή παραδείγματα του πώ η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει πάντα όταν ε, τα κράτη-μέλη δεν σέβονται κατά γράμμα την οδηγία Natura 2000 για παράδειγμα και προκειμένου. Δεν δηλαδή έχουν, ε, δεν έχει αξιολογηθεί το κατά πόσο πληρούνται όλε οι προποθέσει που αναφέρονται στην οδηγία. Και εδώ να σα πω το εξή. Έχουμε, δεν, δεν, έγινε, δεν πληρούνται η προπόθεση για, την ε, για τι σορευτικέ επιπτώσει και κάτι άλλο επίση. Εδώ αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο υπάρχει και είναι σχετική κυκλοφοριακή αλλά θα αυξηθεί πάρα πολύ ε, στο μέλλον. Και δεν εξετάστηκαν και εναλλακτικέ λύσει που υπάρχουν. Αυτό είναι ε, ουσιώδε. Η κυβέρνηση τη Δανία ενέκρινε ένα έργο χωρί να λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία που σα είπα. Ε, υπό το φως όλων αυτών νομίζω ότι η Επιτροπή ε, θα πρέπει ε, να φροντίζει περισσότερο κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, οδηγίες, την οδηγία της συγκεκριμένη, στην προκειμένη περίπτωση. Και ελπίζω ε, να, ε, να, να καταλάβουμε όλοι και να υπερασπιζόμαστε πάντα την αρχή ότι, ε, εάν, ότι έχουμε μια οδηγία που ισχύει. Δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε την οδηγία, αρκεί να σεβόμαστε την οδηγία. δηλαδή, τι νόημα έχει να έχουμε μια οδηγία που ήδη έχει εγκριθεί και να μην μα απασχολεί το κατά πόσο τα κράτη-μέλη, η Δανία στην προκειμένη περίπτωση, σέβονται και πληρούν τι προποθέσει τη οδηγία. Γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το κατά πόσο η οδηγία έχει σεβαστεί όλε τι υποχρεώσει διατάξεις της και έχει τηρήσει όλες τις διατάξεις της οδηγίας. Κοιτάξτε, έχουμε μια έκθεση για την οδηγία ε, Natura 2000 ε, που ακριβώς αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Και να δούμε λοιπόν ποιοι κανόνε δεν γίνονται σεβαστοί. Και καλό την Επιτροπή να ε, αναλάβει, τα, να εκπληρώσει τα καθήκοντά τη που είναι να είναι θεματοφύλακα όλων αυτών των οδηγιών. Δηλαδή, να δεί στην προκειμένη περίπτωση, έγινε μελέτη για τι ορευτικέ επιπτώσεις και εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσει. Αυτά τα δύο πράγματα, κατά την άποψή μου, δεν τηρήθηκαν. Ε, τι προτείνετε λοιπόν, κύριε Όκερ, να, στείλουμε, να, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να, να, να συμπληρώσει την έρευνα όταν την έχει περατώσει. Δεν καταλαβαίνω, επειδή δεν έχω και εμπειρία στι διαδικασίε. τι θα πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να λύσουμε. Γιατί εδώ φαίνεται ότι έχει περατωθεί η έρευνα. Περιμένω από εσά μια πρόταση. Okay, I'll try to do it in English. <laughs> it might be due to the translation. I think that uh, the Commission should... Λοιπόν, θα μιλήσω στα αγγλικά. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή πρέπει όχι μόνο να εξετάσουμε τις επιπτώσεις συγκεκριμένα αυτού του αυτοκινητοδρόμου, αλλά τις σωρευτικές επιπτώσεις στην περιοχή. Όταν δηλαδή αυξάνεται η κυκλοφορία. Έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Εγώ, τώρα τι να σου πω, εγώ θα βρω το πιο, δεν νομίζω ότι εγώ πρέπει να βρω τον πιο κομψό τρόπο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ε, αυτό ε, είναι ανοιχτό σε όλους. Α, είναι πιο εύκολο λοιπόν από ό,τι νόμιζα, γιατί από ό,τι με ενημερώθηκα, ότι η γραμματεία είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να στείλουμε μια επιστολή στην, Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κρατήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή μέχρι να πάρουμε συμπληρωματικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ. στο κομμάτι Straubing-Wilshofen. Ε, Από τη μεριά της ε, Επιτροπής, ε, ο κύριος Τσέζαρε Μπερναβέη. Ο κύριος Τσέζαρε Μπερναβέη. Σας ευχαριστώ. Έχουμε την αναφορά του κυρίου Χούμπερ σε σχέση με με ένα ε, πρόβλημα που έχει να κάνει με την πλωτή οδό ε, του Δούναβη, σε αυτό, εδώ, σε αυτό το τμήμα Στράουμπιν και Βιλσόφιν. Εμείς ε, στα πλαίσια ε, τη βελτίωση όλων των μέσων μεταφορά για να έχουμε ένα υφόρο σύστημα μεταφορών ε, ε, επιβατών και εμπορευμάτων. Και εδώ οι εσωτερικέ πλωτοί οδοί αποτελούν ένα σημαντικό μέρο τη πολιτική μα από μόνε του ή σε συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφορά. Ο Δούναβη, λοιπόν, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορά, έχει προτεραιότητα. Η σε συνδυασμο με αλλα μεσα μεταφορα ο δουναβη λοιπον στα πλαισια των ευρωπαικων δικτυων μεταφορα εχει προτεραιοτητα η ναυσιπλοεια του είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σύνδεση των πλωτών οδών του Βορρά τη Ευρώπη και τη Νότια Ανατολική Ευρώπη. Αλλά ο Δούναβη δεν αποτελεί μόνο ε, μία οδό μεταφοράς, ταυτόχρονα ε, αποτελεί και, με, και, μέρος της περιβαλλοντικής ε, κληρονομιάς και θα πρέπει να το προστατεύουμε. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την κατασκευή του τμήματος μεταξύ των τμήματων αυτών της Βαβαρίας και όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων για την εξασφάλιση της ναυσιπλοείας, για να είναι, για να είναι συμβατές αυτές οι δύο πτυχές, δηλαδή εσωτερική ναυσιπλοεία αλλά και προστασία του περιβάλλοντος προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από τα εμπλεκόμενα μέρη να δημιουργηθεί μια επιτροπή παρακολούθησης η οποία θα παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή τις ε, εργασίες αυτές, ε, θα επαληθεύει ε, την συμμόρφωση με την υφιστάμενη περιβαλλοντολογική νομοθεσία και την χρησιμοποίηση τεχνικών που θα είναι απόλυτα συμβατές. Συμμετείχαν τέσσερα άτομα επιχειρηματίες της Γερμανίας επιφανής και επιφανής περιβαλλοντολογικής περιβαντολόγοι ε, και πρέπει να πούμε ότι ο δόκτωρ Άντων Χούμπερ αποτελεί μέρο τη ομάδα αυτή. Η ομάδα συνήλθε για πρώτη φορά στι 5 Φεβρουαρίου του 2010. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, όσον αφορά ε, ε αυτή την ε, μη, ε, την μία, μία χαρακτήρα, δεν, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι τέτοιο. Η αρχή της συνεργασίας ανάμεσα στους επιχειρηματίες και στους περιβαντολόγους αποτελεί την καλύτερη έκφραση της συμφωνίας που υπέγραψαν οι γειτονικέ χώρες και συμφωνία απόλυτα με τις βασικές αρχές ανάπτυξη εταιρική προστασίας αλλά και της περιβαλλοντικής προστασίας στη λεκάνη απορροής του Δούναβη. Αυτά είχα να πω ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Ε, äh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, επί της ουσίας λέμε ότι στις συμμετέχουσες χώρες λαμβάνει η χώρα τώρα μια συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα του διαδρόμου του, ε, Ο πρώτος περνάει από το Δούναβι και έχει εξαντληθεί ε, η, η δυνατότητα αξιοποίησής του και θα πρέπει να δούμε τι εναλλακτικές υπάρχουν ούτως ώστε να υπάρχει μεταφορική ε, ικανότητα περισσότερη. Η Κομισιόν ε, ανέφερε τα σημαντικότερα, είπε ότι θα παρακολουθήσει τα περαιτέρω και θα απελευθερώσει τα κονδύλια όταν βεβαιωθεί ότι όλες οι περιβαλλοντικές ε, ε, έρευνες έχουν γίνει, διεκτιμήσεις και θα λαμβάνονται υπόψη από το έργο που θα κατασκευαστεί. Οπότε πρέπει να τηρηθεί ανοιχτό το θέμα στην Επιτροπή και όταν πάρουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε δηλαδή την αναφορά αφού δεν έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν μας έχουν αυτές ακόμη διατεθεί. Θα πρέπει λοιπόν να αναμένουμε. Ευχαριστώ όμως την ε, Κομισιόν η οποία ε, επέδειξε συνέπεια και δεν θα ε, προχωρήσει στην χρηματοδότηση πριν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Το κρατάμε λοιπόν ανοιχτό και τηρούμε στάση αναμονής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρη. Uh, is there Ποιος άλλος ε, επιθυμεί να λάβει το λόγο. Γίνεται μια μικρή μετατροπή στην σειρά των ε, επόμενων θεμάτων. Ε, ο αναφέρον κύριος Ανδρέας Βαρνακιώτης της υπόθεσης 22, επειδή θα πρέπει να φύγει σήμερα το βράδυ, παρακαλεί αν είναι δυνατό να μιλήσει πριν από το, αμέσως τώρα πριν από τον αριθμό 20 ε, ο οποίος ευγενικά παραχωρεί ο κύριος Κοκάλας παραχωρεί τη θέση του. Αν συμφωνείτε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαρνακιώτη σχετικά με ένα... Με, με, με, κατασκευή χιτά. Κατασκευή χιτά στην ε, χαΐα της, ε, της Πελοποννήσου. τον κύριο Βαρνακιώτη παρακαλώ. κύριε πρόεδρε της επιτροπής αναφορών κύριε εκπρόσωπε της ευρωπαϊκής επιτροπής κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές μέλη του κοινοβουλίου σας ευχαριστώ που εξετάζετε την αναφορά μου που υπέβαλα και η οποία δεν αφορά εμένα αλλά αφορά 9.500 κατοίκους. Ευχαριστώ επίσης και τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συνοδεύουν την αναφορά μου αυτή και πιστεύουν στο δίκαιο του αιτήματό μας. Επειδή γνωρίζετε ότι μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις, όπως υπόθηκε. Και επειδή δεν έχω χρόνο να σας τις πω τις χίλιες λέξεις, γι' αυτό σας δείχνω τη φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία της θέσεως Παπα-Νικολού, ελαιώνες, αμπελώνες, που θέλουν να κατασκευάσουν χιτά. Επίσης, σας έφερα και τα προϊόντα από την περιοχή αυτή που είναι λάδι και κρασί και σταφίδα για να δείτε πού πάνε να κατασκευάσουν χιτά. Αυτά θα τα δώσω στην Επιτροπή και ευχαριστώ να πιείτε στη συνέχεια ένα ποτηράκι για να δείτε τι βγάζει η περιοχή που θέλουν να την κάνουν νεκροθαφείο σκουπιδιών. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η κατασκευή του χιτά στην περιοχή αυτή είναι παράνομη, είναι αντίθετη με την τεχνολογία, είναι αντιοικονομική, είναι ξεπερασμένη σε εποχής και επιπλέον επικίνδυνη για την υγεία τη δικιά μας, των παιδιών μας και ημών των τουριστών γιατί επισκέπτεστε κατά πολλές χιλιάδες την περιοχή του Κορινθιακού κόλπου. Τώρα θα σας αποδείξω με έγγραφα ότι η κατασκευή κοιτά στην περιοχή Παπα-Νικολού έχει τα στοιχεία αυτά. Νομικά, το δασαρχείο πατρών με το από 7 Οδόου 2003 και με αριθμό πρωτοκόλλου 67-69 όπως έχω καταθέσει τα έγγραφα επάνω και με το από 5 έκτου του 2007 και με αριθμό πρωτοκόλλου 52-79 και σύμφωνα με τον νόμο 3208 του 2003 το δάσος απαγορεύεται να καταστραφεί και να γίνει χιτά εκτός από δάσος όπως χαρακτηρίζεται η μισή τουλάχιστον περιοχή η υπόλοιπη χαρακτηρίζεται από αγροτικές εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας και ελαιοκαλλιέργειας. Από εκεί είναι και τα μπουκάλια που σας έφερα, από εκεί είναι και το δείγμα αυτό. Δεύτερον, η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Με το από 13 Πέμπτου 2009 έγγραφο και με αριθμό πρωτοκόλλου 2433 προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στέλνει αναφορά των κατοίκων της περιοχής Μυρόδρυσης όπου και ανήκει διοικητικά η Παπανικολού και στέλνει ειδικά την ένσταση της κατοίκου Βασιλικής Γεωργίου Ρούσου γιατί διαμαρτύρεται. Ζητά την βεβαίωση χρηματοδότηση του έργου για την περιφέρεια Δυτική Ελλάδο, ισχυρίζεται πω την έχει, μέχρι σήμερα δεν έχει πάει. Παρακαλεί να τη απαντήσουν ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία και απάντηση δεν έχει πάρει Α σημειωθεί την περιφέρεια κάνει δημοπράτηση χωρί προηγουμένω να έχει κάνει απαλωτρίωση. Δεν έχει γίνει απαλωτρίωση στην περιοχή. Επιπλέον, επειδή ο χρόνο είναι ελάχιστο και τον σέβομαι για η κούρασή σα μεγάλη, επιπλέον θέλω να σα πω ότι στην περιοχή μα υπάρχουν τρεις που λειτουργούν. Οι τρεις χιτά είναι ικανοί να καλύψουν τα σκουπίδια αυτή τη συγκεκριμένη ενότητα που μιλάμε. Σε δύο χρόνια κατασκευάζεται δε εργοστάσιο επεξεργασίας σκουπιδιών που θα μας υποχρεώσουν να πάμε τα σκουπίδια εκεί. Προς τι λοιπόν αυτή η σπατάλη των 7 εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή που η χώρα μας όπως και η Ευρώπη έχει οικονομικό πρόβλημα και ο Πρωθυπουργό μας γυρίζει για να μπορέσει να περισσώσει κάποια κονδύλια. Εμείς θα πάμε να σπαταλήσουμε 7 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν υπάρχει λόγος. Πιθανόν μερικοί να πούν ότι εγώ αντιτίθεμαι στην πατρίδα μου. Δεν είναι έτσι. Προσπαθώ να προφυλάξω από λάθη τα οποία έχουν ξεκινήσει από καιρό. Δεν είναι σημερινά. Τα λάθη λοιπόν αυτά ήθαμε να, τα βοηθήσετε, να μας βοηθήσετε να τα αποφύγουμε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, για να μην σα κουράσω, έχω καταθέσει τα έγγραφα. Ο νόμο 1650 από τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 12, 18, 19, 22 και 28 που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος όπως και στην περιοχή Natura που ανήκει η περιοχή δική μας που έχει νερά όπως λέμε από εκεί πίνουμε νερό έχει 248 γεωτρήσεις από εκεί πίνουν 12 διαμερίσματα νερό ε, αταγνοούν αυτά όλα και την υδροδότηση του ποταμού αλλά και την υδροδότηση που παίρνουμε από τις 248 γεωτρήσεις λυπηθείτε μας πλέον θα πεθάνουμε δεν έχουμε άλλη δυνατότητα αυτός λοιπόν ο χώρος έχουν επιλέξει για να τον κάνουν χιτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εσείς αν ήσασταν στη θέση μας τι θα κάνατε. Τώρα με αυτά που σας είπα δεν ακούτε τη φωνή μου. Δεν μιλάω εγώ. Ακούτε τη φωνή 9.500 κατοίκων. Ακούτε τη φωνή των παιδιών μας, τη φωνή των μεγαλύτερων μας που μας κοιτάζουν διαρκώς με κραμμένα μάτια και χίλιοι που ψελίζουν και λένε «Λοιπόν η Ευρώπη θα μας αφήσει να πεθάνουμε» αυτό το παράπονο μου είπα να σας μεταφέρω και σας ρωτάω κυρίες και κύριοι βουλευτές της Ευρώπης εσείς που έχετε ιστορικά συνδεθεί με τον τόπο μας μέσα από τόσε δίκαιε αντιδράσει, επαναστάσει και πολιτιστικέ δόξες όπω έγινε με τον Κάρολο τον Μέγα, τον Όθανα τον Πρώτο, με του Γάλλου διαφωτιστέ και με τον ομφάλιο λόρο που συνδέει πολιτιστικά την κλασική Ελλάδα με τη Ρώμη. Μην μα αφήσετε στο έλεο κάποιων παραλογισμών. Τον φιλελληνισμό σα τον ξέρουμε, τον έχετε δείξει πάρα πολλέ φορέ και ειδικά όταν ήταν κλεισμένο το μεσολόγιο έτοιμο να πεθάνει. Και εμείς εγμαλωτισμένοι νιώθουμε. Δώστε μας το δίκαιο μας και την απελευθερωσή μας. Αποχαιρετώντα σας, ρωτώ την ανθρωπιά σας, τον πολιτισμό σας, το αίσθημα του δικαίου και της ένωσης που έχουμε. Κάνω έκκληση σε αυτά. Θα μας εγκαταλείψετε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Βαρνακιώτη. Ε από τη μεριά της Επιτροπής ο κύριος Κουνινιώτης. Είναι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση των ονομάτων. Ε, και με αν μια κατάληξη, ότις ότις. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ναι, όντως έχουμε και και οικογένεια εκεί πέρα. Ε, λοιπόν, σύμφωνα με τον αναφέρον, ο ελόγο χώρο υγειονομική ταφή αποβλήτων προβλέπεται να κατασκευαστεί χωρί κοινωνική συνένεση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, κοντά σε αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία και κατά μήκο του ποταμού Φίνικα, ο οποίο σε απόσταση μόλι 6 χιλιόμετρων εκβάλλει στη θάλασσα. Επιπροσθέτω, σύμφωνα πάντα με τον αναφέρον, η περιοχή είναι σεισμογενή. Η παρούσα αναφορά είχε πρόσφατα αρχαιοθετηθεί από την Επιτροπή Αναφορών, αλλά βάσει νέων στοιχείων η Επιτροπή σα έλαβε την απόφαση να την ξανανοίξει. Πιο συγκεκριμένα, ο αναφέρον απέστειλε μια μελέτη που έγινε <clears throat> από μια ανεξάρτητη εταιρεία εμπειρογνώμων και που καταλήγει στην ακαταλληλότητα τη θέση που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του χώρου υγειονομική ταφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αναφέρον είχε επίση αποστέλει καταγγελία στην Επιτροπή, η οποία του είχε απαντήσει στι 11 Ιουλίου 2007 και του είχε ζητήσει να τη στείλει νέα στοιχεία ικανά να αποδείξουν την ύπαρξη παράβαση τη κοινοτική νομοθεσία ο καταγγέλων δεν είχε τότε απαντήσει στην επιστολή της Επιτροπής. Μετά την ανάλυση της ε, εν λόγω μελέτης που απέστειλε, η Επιτροπή θα ήθελε να ξανά επιβεβαιώσει την αρχική της θέση που είχε ήδη εκφράσει την Επιτροπή Αναφορών και να καταλήξει στην μια παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον για τους λόγους που θα σας αναφέρουμε. Η Επιτροπή θα ήθελε αρχικά να διευκρινίσει ότι η υγειονομική ταφή αποβλήτων δεν απαγορεύεται <clears throat> από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά αποτελεί μια επιτρεπόμενη μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την Οδηγία 9931 για τα απόβλητα. Η κατασκευή χώρων διάθεση αποβλήτων πρέπει να υποβληθεί σε άδεια και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία 85 85-347, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επηρεάσει την απόφαση των εθνικών αρχών Ω προ τη σκοπιμότητα κατασκευή και την χωροθέτηση ενός έργου ή να προβεί σε έλεγχο ουσία της μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των <clears throat> εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Όλα αυτά αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών. Η μόνη εξαίρεση που υπάρχει σε αυτόν τον κανόνα είναι οι περιπτώσει όπου το κράτο μέλο υποπίπτει σε πρόδειλο σφάλμα εκτιμήσεω. Ωστόσο, η ύπαρξη και μόνο μια μελέτη από ανεξάρτητου επιδογνώμονε, η οποία βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν αποτελεί ένα τέτοιο πρόβλημα σφάλμα εκτιμήσεω. Η Επιτροπή θα ήθελε επίση να προσθέσει ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν περιέχει διατάξει σχετικά με τι ελάχιστε αποστάσει μεταξύ των χώρων υγειονομική ταυτή αποβλήτων και την θάλασσα, των αρχαιολογικών μνημείων, τι δασικέ εκτάσει ή τι σεσμογενεί περιοχέ. Η χωροθέτηση των εν λόγω έργων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Θα πρέπει επίση να επισημαθεί ότι δυνάμει τη Οδηγία 2006-12 η απόφαση για το επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή νομαχιακό του σχεδιασμού διαχείριση αποβλήτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, στην διακριτική ευχαιρεια των οποίων ανήκει και η επιλογή των μεθόδων και των χώρων διάθεση. Όλα αυτά δεν μπορούν να <clears throat> αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από την Επιτροπή. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ελληνικέ αρχέ, στα πλαίσια συμμόρφωση με τι διατάξει τη οδηγία αυτή, έχουν υιοθετήσει το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο με διάφορε κοινέ υπουργικέ αποφάσει. Πρέπει επίση να τονιστεί ότι η Οδηγία 85347 περιέχει όντω διατάξει σχετικά με την ενημέρωση του κοινού σε αρχικό στάδιο των διαδικασιών λήψη αποφάσεων και την δυνατότητα να συμμετάσχει στι διαδικασίε λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, αν και οι εθνικέ αρχέ πρέπει να λάβουν υπόψη τι παρατηρήσει και γνώμε που εκφράστηκαν από το κοινό, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση βάσει τη κοινοτική νομοθεσία να τι ακολουθήσουν. Όσον αφορά, τι <clears throat> αφορά τις αιτιάσεις του αναφέρον ότι η κατασκευή και η λειτουργία του εν λόγω χώρου υγειονομική ταφή αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον, όπως π.χ. η ρήπανση των υδάτων, η ενδεχόμενη παραβίαση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα και τα ύδατα θα εξαρτηθεί από το αν ο χώρο θα λειτουργήσει σύμφωνα με τι διαγραφέ και τι διατάξει τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σα ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι γνωρίζω τον αναφέροντα, τον γνωρίζω διότι έχει έντονη κοινωνική δράση στην Ελλάδα, πλέον της ιδιότητάς του ως δημάρχου του Δήμου Ερηναίου. Ε, πέραν όμως της αναφοράς του ε, αναφέροντος, έχω στα χέρια μου επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με το συγκεκριμένο έργο και από άλλους οκτώ δημάρχους της περιοχής και επίσης έχω μια άποψη σχετικά με την περιοχή η οποία ε, είναι η αυτή με τον αναφέροντα. Δηλαδή, ο τόπος ο οποίος έχει επιλεγεί για να γίνει ο συγκεκριμένος χιτάρ είναι πολύ κοντά ε, σε ένα ποταμό ο οποίος λέγεται Φινίξ και ο οποίος είναι ποταμός ο οποίος αρδεύει την περιοχή και από τον ποταμό αυτό εξαρτώνται όλες οι καλλιέργειες, οι γεωρικές καλλιέργειες της περιοχής Πλέον δε τούτου υπάρχουν και διάφορες ε, ε διανοίξεις πηγαδιών από τις οποίες ιδρεύεται η περιοχή. Συνεπώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από την τοποθεσία στην οποία ε, σκοπεύει δια της υπουργικής, ε, αποφάσεως αυτής που προσβάλλεται του γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργηθεί πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα με τα συνεπακόλουθα και στις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και στην υγεία των ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή και υπερβαίνουν τους 10.000. Ε, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ε, αναφέρεται ε, ο κύριος ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο οποίος εξ ονόματος φαίνεται να κατάγεται και από εκείνη την περιοχή της Κορινθίας, από μια διπλανή περιοχή, ε, δεν αναφέρεται αν πράγματι υπάρχει ΕΠΕ για το συγκεκριμένο θέμα και οδηγία για τα ύδατα, διότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίες για τα ύδατα εν προκειμένου, που συνδέεται αρρήκτως με τη ζωή των προσώπων. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε με πολύ σοβαρότητα το θέμα και να ζητήσουμε διευκρινήσεις πολύ δε περισσότερο όταν κατά την άποψή μου υπάρχει σπατάλη 7 εκατομμυρίων, όχι επειδή τα βρήκαμε τα 7 εκατομμύρια έτσι εύκολα να τα πετάμε και, πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα διότι οι τοπικοί παραγόντες έχουν πιστέψει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ταμείο το οποίο μοιράζει λεφτά. Λοιπόν, δεν πρέπει να μοιράζει λεφτά, πρέπει να μοιράζει ωφέλιμα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα οποία μοιράζει πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένου σκοπούς και να εξυπηρετούν τους σκοπούς με βάση την ωφελημότητα. Λοιπόν, ε, σε δύο χρόνια, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα έχει δημιουργηθεί ένα μείζον έργο το οποίο θα επικαλύπτει και θα καλύπτει τις ανάγκες. Επομένως εγώ θεωρώ ω γνώση τη περιοχή ότι τα 7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χρηματοδοτούμε από την κοινότητα θα πάνε στον αέρα. Και παρακαλώ πάρα πολύ να το λάβετε αυτό πολύ σοβαρά υπόψη, να το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα και να ζητήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση διευκρινήσει, ιδιαίτερα με, την, ε, με τον συνδυασμό του εάν και κατά πόσον είναι απαραίτητο ο χιτά αυτός να γίνει εν ώψη του γεγονότος ότι ήδη ολοκληρώνεται μια άλλη διαργασία, πώς την είπατε, κατασκευή εργοστασίου αυτού στην ίδια περιοχή. Θέλουμε απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Επιτροπή να ζητήσει άμεση απάντηση εάν καλύπτονται οι ανάγκε τη περιοχή από το ήδη υποκατασκευή άλλο έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Έτσι. Ε, θέλετε να στείλει επιστολή η Επιτροπή. Να Επιτροπή ε, στην οποία να λέει ότι πληροφορηθήκαμε ότι στην περιοχή σας δημιουργείται ένα έργο που θα καλύψει τις ανάγκε ανάγκες των κατοίκων από πλευράς αποβλήτων και το οποίο ολοκληρώνεται εντός των προσεχών μηνών. Να συνδυαστεί το έργο αυτό, εάν και κατά πόσον έχει το capacity να καλύψει την, ε, της περιοχής της ανάγκης τρόπον ώστε να μην πεταχτούν αφενός να μην πεταχτούν 7 εκατομμύρια ευρώ αφετέρου να μην δημιουργήσουμε κοινωνική αναταραχή. Πολύ σας ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Γιάρ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Η χιτά πάντα ε, έχουν ένα στοιχείο επικίνδυνοτητας που περνάει στην επόμενη γενιά. Και στη Γερμανία, την Ανατολική Γερμανία, στα Ανατολικά κρατήδια, ε, είχαμε κάποιες ε, κληρονομιές από το πρώην σοσιαλιστικό καθεστώς που έπρεπε να λύσουμε και να ξεπεράσουμε. Δηλαδή είναι αυτό το ζήτημα των χωματερών είναι ένα θέμα που πρέπει να το βλέπουμε πολύ προσεκτικά. Ε, η Κομισιόν, όπως την ακούσαμε, είπε ότι αφενός δεν μπορεί να παρέμβει εκτός και αν υπάρξουν σαφή ε, λάθη αξιολόγησης. Ε, αν δούμε εδώ τον οικισμό που είναι κοντά, αν δούμε τον ποταμό που είναι στην άμεση, σε άμεση γυτνίαση, ε, δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Είναι, υπάρχουν ανοιχτά θέματα που συνηγορούν υπέρ του να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και να απευθύνουμε και μία επιστολή που θα επισημαίνει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα εδώ. Άρα νομίζω ότι πρέπει να παρεμβούμε. Συμφωνώ δηλαδή εδώ με τους προλαλήσαντες. Δεν ξέρω ε, αν μπορούμε να, επι... επιβάλλουμε στις ελληνικές αρχές τι είναι σόφρον και σωστό και τι όχι. Ε, αλλά νομίζω ότι και η Κομισιόν, αν την ερμήνευσα καλά, είπε ότι ε, θα πρέπει να προϋποθέσουμε ότι οι αρχές κινούνται σωστά, αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε εάν εξήτασαν το θέμα στο εύρος που θα άξιζε να εξεταστεί το θέμα. Μπορούμε να το πούμε και αυτό και ίσως να συμπεριλάβουμε και μια έκκληση που θα λέει ότι σήμερα υπάρχουν πιο έξυπνες μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης των απορριμμάτων από το να τις καταχώνουμε, τα, καταχώνουμε κάπου. Σχολιάσω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική στροφή στην ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα τον τελευταία, τελευταίους μήνες με την έννοια ότι πολλά, πολλές από αυτές τις αποφάσεις που πάρθηκαν παλαιότερα επανεκτιμώνται Επομένως είναι πιθανότατα, είναι πολύ σημαντικό να σταλεί αυτή η επιστολή και να ενημερωθεί για το ενδεχόμενο και να μας απαντήσει για τα σχέδια. ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας. Κυρία Μπελιέ. Θα κινηθώ και εγώ προς την ίδια κατεύθυνση με τους προλαλήσαντες συναδέλφους ένα στοιχείο στην ε, απάντηση της Κομισιόν ε, μου δημιούργησε επιφυλάξεις όσον αφορά τον αντίκτυπο στο νερό. Μας λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο εξαρτάται από τον αντίκτυπο στο νερό και μας λένε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση που να μας δείχνει ποιος ακριβώς θα είναι ο αντίκτυπος στο νερό. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκτιμήσεις που θα μας διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει αρνητική επίπτωση στο νερό. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν κίνδυνοι και έχουμε μπροστά μας αυτή την αναφορά, άρα πρέπει εμείς να ενημερώσουμε την ελληνικές αρχές ότι υπάρχει ανεπάρκεια όσον αφορά το θέμα της ενημέρωσης για τις επιπτώσεις. Κυρία Γιώτοβα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τα επιχειρήματα του αναφερόντος καθώς και με τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από εμένα. Νομίζω ότι πρόκειται για θέμα όπου δεν πρέπει να παραμείνουμε αμερόληπτοι και αντικειμενική. Θα έπρεπε να στείλουμε μία επιστολή στις αρχές και ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες θα μπορούσαμε να στείλουμε επιτόπου μία μικρή αποσταλή για να διαπιστώσουμε αν όντως υπάρχει η παραβίαση της οδηγίας ή όχι. Να πω ότι έχουν προσπαθήσει πολλές φορές οι ελληνικές αρχές να φτιάξουν χωματερές και όντως εδώ πρόκειται για περίπτωση όπου θα έπρεπε να έχουμε μια επιτόπου επίσκεψη. Ε, απλώς να προσθέσω, από ό,τι έχω, από ό,τι μάθει, η υπόθεση αυτή έχει πάει επίσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, οπότε ίσως να είναι και σοφό να περιμένουμε να δούμε και αυτή η Εθνική Δικαιοσύνη τι θα αποφασίσει, γιατί όπως ξέρετε ο Εθνικός Δικαστής ε, ε, έχει και το, την, την ικανότητα να εφαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο εννοείται να περιμένουμε να απαντήσουμε στην ελληνική, να διευκρινίσουμε ζητήματα από την ελληνική κυβέρνηση μέχρι ότου βγει το όχι. Δεν ξέρω πότε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία αναμένεται. Το ένα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το άλλο. Ε, Επομένω, γράφουμε ένα γράμμα. Ε, κύριε Βοστινάρου, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ. Όχι αντίρρηση. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο σχόλιο. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, οδηγίες, κανονισμοί. Και όλα μοιάζουν τέλεια. Όμως, όταν φτάνουμε στην εφαρμογή των κανόνων αυτών, διαπιστώνουμε ξαφνικά ότι τα κράτη-μέλη είτε αποτυγχάνουν στην εφαρμογή των κανόνων που υπάρχουν ή κάνουν πολύ κακή ελλειπή ερμηνεία των κανόνων αυτών. Και εδώ επανέρχομαι στην έκθεσή μου για τη βιοπικιλότητα. Το ίδιο πράγμα, το έχουμε ξαναδεί. Αποτυχία των κρατών μελών να εφαρμόσουν σωστά τις οδηγίες. Και επίσης μία πραγματικά απαράδεκτη στάση των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιμένουν, που αφήνουν στις καλένδες τις επίσημες απαντήσεις. Πρώτα απάντηση από την Εθνική Κυβέρνηση, μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μεταξύ είτε προχωράνε τα έργα αυτά και ορισμένες φορές δημιουργούν ανήκες στο βλάβη είτε ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι δεν προστατεύονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αποτυγχάνει λοιπόν στον θεσμικό της ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να ζητάμε πάντα ταχείες απαντήσεις από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να μην περιμένουμε παέριστο. Επίσης, αντιδράσεις άμεσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος πρέπει να ζητάμε και σωστή εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων από τις εθνικές κυβερνήσεις. Αν δεν το κατορθώσουμε αυτό, θα αποτύχουμε δραματικά στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί είμαστε συνεργοί πλέον και είμαστε υπεύθυνοι εφόσον δεν αντιδρούμε και εφόσον δεν ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να συμπεριφέρονται σωστά. Το πρόβλημα δεν είναι οι κανόνες και οι κανονισμοί, είναι η εφαρμογή τους. Και αυτό το πρόβλημα δεν θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτό. Ξεκινήσαμε το 2007, τώρα είμαστε αρχές 2012 και ακόμη περιμένουμε από τα τοπικά συμβούλια να απαντήσουν, από το Συμβούλιο Επικρατείας να απαντήσει και τελικά παραπέμπουμε τα πάντα στις καλένδες. Νομίζω ότι καταλάβατε πολύ καλά τις προθέσεις μου, κυρία Παλιαδέλη. Κυρία Πρόεδρε, να παρακαλέσω κάτι, αν τελειώσαμε με το θέμα επειδή πρέπει να φύγω για την Αθήνα, ε, παρακαλώ, το 20 θέμα είναι αίτημα του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είναι βουλευτής του κόμματός μας και δεν μπορεί να παραστεί διότι υπάρχουν αλληλημένες υποχρεώσεις και ψηφοφορίες που ξέρετε κάτω. Και εγώ φεύγω σήμερα για να είμαι σε μια press conference για τα οικονομικά μεθαύριο. Η παράκληση είναι να αναβληθεί η εξέταση του θέματος για ευθετότερο χρόνο, παρακαλώ. Δεν μπορούσε να έρθει οπωσδήποτε. Uh, uh, Στο 21 αναφέρεστε. Ο αναφερόμενος είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ζητάει αναβολή της εξέτασης προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί. Εντάξει, για το σημείο 21. Ωραία. Τώρα περνάμε στο σημείο 20. Και παραβρίσκεται ο κύριος Κοκάλας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Την αναφορά 669 του 2006 για την παράνομη και ανεξέλεγκτη χωματερή των σπετσών, στην οποία πετιούνται αδιακρίτως όλα τα απόβλητα του νησιού, δεν την υπέβαλα μόνον εγώ, υπογράφουν και δύο επιφανείς ε, πρέσβεις της Ελλάδας που κατοικούν στο νησί και επιπλέον έχω την άδεια να σας μεταφέρω και τη μαρτυρία του Προέδρου της Βελγικής Γερουσίας, του κυρίου Αρμάν Ντεντεκέρ, που το περασμένο καλοκαίρι δεν πίστευε στα μάτια του όταν αντίκρισε το θέαμα της χωματερής αυτής. Οι Σπέτσες ε, κατοικούνται το χειμώνα από 6.000 περίπου μόνιμους κατοίκους τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά από τον εσωτερικό τουρισμό και από τις χιλιάδες Αθηναίους που έχουν φτιάξει εκεί τις ε, εξωγικές τους κατοικίες, τις οποίες επισκέπτονται σε μόνιμη βάση. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν εκδοθεί πάνω από 500 άδειες οικοδομής και ότι κατά, κατά την τουριστική περίοδο οι κάτοικοι φτάνουν τις 25.000. Από το 2006 που υπευλήθη η αναφορά, η κατάσταση στις Πέτσες έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Η εν λόγω παράνομη χωματερή θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη στην Ανατολική Πελοπόννησο. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές χωματερές. Καμία καμία, το επαναλαμβάνω, δεν ρηπαίνει τη θάλασσα και τον αέρα όσο η συγκεκριμένη. Και αυτό γιατί βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη θάλασσα, σε ένα εντελώς απροστάτευτο από τους ανέμους και τις βροχές σημείο. Με κάθε δυνατή βροχή ξεπλένεται ένας τεράστιος όγκος σκουπιδιών, κάθε είδους, και τα αποστραγγίσματα καταλήγουν στη θάλασσα. Με κάθε ρηπή ανέμου ο καπνός και τα δηλητηριώδη αέρια που παράγονται από τη μόνιμη, μόνιμη φωτιά που καίει τα πλαστικά και τα οργανικά υλικά μεταφέρεται χιλιόμετρα μακριά και δεκάδες σακούλες και χαρτιά πετούν στον αέρα. Όλα αυτά καταλήγουν πάλι στη θάλασσα. Η χωματερία αυτή τροφοδοτεί με σκουπίδια όλες τις ακτές της Ανατολικής Πελοποννήσου. Και από αυτήν έχουν ξεκινήσει δύο μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κατακάψει ένα σπάνιας πυκνότητας πευκοδάσος. Στο ίδιο σημείο της κομματερής ρίχνονται από και τα λίματα των σπιτιών, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων του νησιού. Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, όλοι εξυπηρετούνται από βιτία. Η τοπική αρχή ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να κατασκευαστεί βιολογικός καθαρισμός και φυσικά λέει ψέματα προτιμάει τα έργα βιτρίνας και πρόσφατα μάλιστα διέθεσε 4.284.000 ευρώ και αναδιαμόρφωσε την κύρια πλατεία του νησιού, περίπου τριών στρεμάτων. Το 80% από τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε πλατεία δεν χρειαζόταν καμία αναδιαμόρφωση ήταν ε, πολύ καλά στρωμένη με τσιμέντο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να καλυφθεί από πανάκριβες μαρμάρινες πλάκες που σε λίγο καιρό θα σπάσουν από το βάρος των διερχόμενων φορτηγών. Και χρήματα συνεπώς υπήρχαν και χώρος για την κατασκευή ενός σταθμού επεξεργασίας των λιμάτων που μεταφέρονται με τα βιτία. Πιστεύω ότι το αποχετευτικό δίκτυο θα μπορούσε να περιμένει να γίνει αργότερα. Για τα σκουπίδια ε, γνωρίζω εδώ και χρόνια ότι υπάρχει ένα σχέδιο να μεταφέρονται σε έναν κεντρικό χώρο υγειονομικής ταφής, στην Πελοπόννησο, έξω από τις Πέτσες, στο Άργος ή στο Ναύπλιο, αλλά ούτε αυτό γίνεται. Στο σημείο αυτό πρέπει να πω δυστυχώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ιδία γνώση για τη σοβαρότητα της κατάστασης και το μέγεθος της μόλυνσης που προκαλεί η εν λόγω χωματερή. Τα στοιχεία μάλιστα που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης δεν είναι αληθινά. Λόγω της ε, πολύχρονης ενασχόλησής μου με σπορ της θάλασσας, γνωρίζω την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου σαν το σπίτι μου. Πιθανή προς πιθανή. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι η ρήπανση τόσο από τα σκουπίδια όσο και από τον καπνό και τα λίματα είναι αισθητή σε μια τεράστια έκταση. Κυρία Πρόεδρε, η θάλασσα από τις Πέτσες έως ε, το νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου, όποιος την διαβεί, κάθε 100-200 μέτρα θα συναντήσει σακούλες να επιπλέουν. Και άλλα επιπλέοντα υλικά. Κάθε λογής επιπλέοντα υλικά. Ο βυθός δε, όχι μόνο στις πέτσες, αλλά και σε τεράστια απόσταση από εκεί, καλύπτεται από ένα είδος σκόνης. Και είμαι βέβαιος ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα επιπλέοντα σκουπίδια και από αυτή τη σκόνη, από αυτό το ίζημα που κάθεται στο βυθό, ακόμη και στην απέναντι ακτή της Πελοποννήσου που απέχει 14 μίλια, ε, σε μια ακτή που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη, δηλαδή δεν ρίχνονται άλλα απόβλητα, έτσι, ε, ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ίζημα αυτό προέρχεται από τις πέτσες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Κοκάλα, παρόλο που για μια Ελληνίδα πρόεδρο είναι πραγματικά ε, τουλάχιστον αμήχανη στιγμή να ακούει και να βλέπει τέτοια πράγματα. Να δηλώσω εξ αρχής ότι πλήρη ευθύνη έχει ο Δήμος Σπετζών φαντάζομαι. Ε, επομένως να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα δούμε όμως τι έχει να μας πει προηγουμένως η, ο εκπρόσωπος του, της Επιτροπής, ο κύριος Μπλέχ. Ε, Mr. I would very much appreciate your opinion. Κύριε Μπλέχ, θα ήθελα την άποψή σας για το θέμα αυτό. Mr. Μπλεχ Thank you, Mrs. Chair. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το σοβαρό της κατάστασης όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων, στερεών αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Με βάση το άρθρο 260 της συνθήκης, πρώην άρθρο 228, κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει για δεύτερη φορά στο δικαστήριο ζητώντας πρόστιμα. Θεωρώ θα ήταν καλύτερο να δοθούν αυτά τα χρήματα για την διαχείριση των αποβλήτων αλλά η ευρωπαϊκή κυβέρνηση, η ελληνική με συγχωρείτε κυβέρνηση προτιμά να τα δίνει για πληρωμή προστήμων. Για την ε, εφαρμογή της απόφασης λοιπόν του δικαστηρίου έχουμε ξεκινήσει ως επιτροπή διαδικασία με βάση το άρθρο 260 της συνθήκης κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εφάπαξη μηνιαίο πρόστιμα. Όσον αφορά τα ύδατα κολύμβησης καταλαβαίνω τον ε, αναφέροντα που μας λέει ότι είναι πραγματικά απέσιο το να βλέπει κανείς πλαστικές σακούλες εκεί που κολυμπάει. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ε, διατάξεις που ισχύουν για τα νερά κολύμβησης, πρέπει να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν κυρίως ε, την μικροβιολογική σύνθεση και τους οργανισμούς που έχουν και άμεση επίπτωση. Άρα δεν μπορούμε αυτό να το κρίνουμε από την ύπαρξη πλαστικών σακουλών, αλλά βεβαίως ε, κάτι τέτοιο ίσως να είναι ένας λόγος για να θεωρήσουμε ότι και η μικροβιολογική κατάσταση δεν είναι καλή. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι αν λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων θα λυθεί και το πρόβλημα των υδάτων κολύμβησης γιατί προφανώς πρόκειται για θέμα που έχει να κάνει με την κατεύθυνση του ανέμου και το πώς τα απόβλητα καταλήγουν στα νερά κολύμβησης. Άλλα σχόλια. Ο κύριος Ποστινάρο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, η κατάστασή μου ε, τώρα είναι πολύ δύσκολη γιατί εδώ δεν συζητάμε μία αναφορά που συνυπογράφεται και από ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ένα μέλος ενός πολιτικού κόμματος. Δεν πρόκειται δηλαδή για πολιτική αναφορά, αλλά πρόκειται για μία αναφορά που αφορά ένα θέμα που το γνωρίζει και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2006. Από το 2006 και μετά ακούμε μόνο εξηγήσεις γιατί δεν έχει εφαρμοστεί κάτι. Και έχουμε ένα πινκ-πονγκ μεταξύ Βρυξελών και Αθήνας που συνεχίζεται και ταυτόχρονα η μόλυνση που η μόλυνση δεν αφορά μόνο τα στερεά απόβλητα αλλά και οργανικές ενώσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί χρειάζονται κάπου 100 χρόνια αν δεν κάνω λάθος προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάσταση των υπογείων υδάτων. Και ενώ συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, εμείς ακούμε μόνο εξηγήσει. Στρέφομαι προς την Επιτροπή. Πώς μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Μας λένε ότι ναι, παραβιάζουν. Μας λένε ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις οδηγίες, ότι έχουν τη θέληση να κάνουν κάτι, αλλά Μόνο αυτό. Μόνο αδύναμες εξηγήσει. Τι θα γίνει με την εφαρμογή, την εφαρμογή των συμπερασμάτων. Αν δεν γίνει αυτό, τότε απλά έχουμε κοινωνικές εκδηλώσεις, κοινωνικές επαφές μεταξύ Κομισιών και Ελληνικής Κυβέρνησης. Αυτή η κατάσταση καταστρέφει την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα, στις Πέτσες, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Γκρινή, ευχαριστώ πολύ. Και εμένα με εκπλήσει καταρχάς το πόσο καιρός έχει περάσει και το ότι συνεχίζει να περνάει ο καιρός. Γιατί είναι πραγματικά τρομακτική η κατάσταση με τις ε, χωματερές αυτή τη στιγμή. Βλέπω την κατάσταση των υδάτων για το 2009 στην Ευρώπη και βλέπω τα στοιχεία για την Ελλάδα. Αναφέρεται εδώ την ποιότητα των υδάτων κολύμβασης. Ενδεχομένως όμως θα ήταν ενδιαφέρον να είχαμε και στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, ελληνικές αρχές, είναι ανησυχητικό το θέμα, γιατί για τους Γάλλους είναι ονειρικός προορισμός η Ελλάδα και ονειρευόμαστε να πάμε στην Ελλάδα για διακοπές. Εγώ σήμερα σκέφτομαι να μην πάω στην Ελλάδα. Ελπίζω λοιπόν τόσο χάρη του πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού, όσο και για εμάς τους τουρίστες ότι θα κάνει κάτι παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι και εμείς η δική μας Επιτροπή θα προσπαθήσουμε να επιμείνουμε προκειμένου να μην επανέλθει σε τρία χρόνια από τώρα ξανά το ίδιο θέμα στην Επιτροπή Αναφορών. I, ναι. I, was really... Ε, ήμουνα και εγώ έτσι, ενοχλήθηκα πάρα πολύ με την εικόνα σε ένα πολύ όμορφο νησί που έχει και ιστορική διάσταση. Δεν είναι απλά ότι είναι στην Ανατολική Πελοπόννησο, είναι συνδεδεμένο και με τη σχετικά νεότερη ιστορία μας, ε, την ελληνική εννοώ. Ε, θεωρώ ότι ε, όταν λέμε ελληνικό κράτος, δεν θα ήθελα να το γενικεύουμε τόσο πολύ, σας παρακαλώ. Περάσαμε και περνάμε μια δύσκολη περίοδο. βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον, με τον τεράστιο αγώνα που κάνει μια νέα κυβέρνηση από τον Νοέμβρη να βάλει τα πράγματα στην θέση τους ε, και να αποκαταστήσει τη σχέση των Ελλήνων πολιτών με την εφαρμογή των νόμων. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια πραγματικά είχε φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτή η έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη εφαρμογής των νόμων. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι λοιπόν όχι γενικώ με ένα ελληνικό κράτος έτσι, το οποίο είναι υπεύθυνο, αλλά με μια κυβέρνηση που αυτόν τον καιρό προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ θα ενημερώσω αμέσως, ήδη προσπάθησα να το κάνω σήμερα το πρωί, αλλά προτείνω να κάνουμε το εξής, να γράψουμε ένα πολύ αυστηρό γράμμα στον Δήμο που, υπάγεται, που κάνει αυτό το έγκλημα, το οποίο να κοινοποιήσουμε στην ελληνική κυβέρνηση και να παρακαλέσουμε την Επιτροπή παράλληλα να συνεχίσει να πιέζει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 Τώρα έχουμε ένα άλλο ελληνικό θέμα του κυρίου Παναγιώτη Μπούρα. Ο κύριος Κουνινιώτη πάλι θα παρουσιάσει το ζήτημα. Η αξιολόγηση της παρούσα αναφοράς από την Επιτροπή αφορά την ενδεχόμενη παραβίαση όχι μόνο της οδηγίας 9931 και τα απόβλητα, αλλά και τις οδηγία 85347 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ερωτησμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97-11 και 2003-35. Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου η Οδηγία 9931 μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο προβλέπει την έκδοση απόφαση έγκριση των περιβαλλοντικών όρων πριν από την υποβολή ε, αίτηση για την χορήγηση άδεια λειτουργία χώρου υγειονομική ταφή από τον φορέα εκμετάλλευση η απόφαση έκδηση των περιβαλλοντικών όρων χορηγείται σύμφωνα με τι διατάξει δια των οποίων μεταφέρεται η Οδηγία 85-337 ΕΟΚ στο ελληνικό δίκαιο. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι κινήθηκε η διαδικασία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω έργου στο περιβάλλον. Ειδικότερα, <clears throat> ειδικότερα ο αρμόδιο Υπουργό ενέκρινε προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου. Εν τούτης, η έγκριση της συγκεκριμένη πράξης συνιστά μόνο προκαταρτικό στάδιο και δεν παράγει δευμεστικά ένομα αποτελέσματα. Πράγματι, ο κύριος του έργου <clears throat> οφείλει να εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία τίθεται εν συνέχεια στη διάθεση του κοινού και των αρχών που ενδέχεται να εμπλέκονται. Κατόπιν, η αρμόδια αρχή πρέπει να προβεί στη λήψη τελικής απόφασης. Δεδομένου ότι η διαδικασία εκτίμηση και χορήγηση άδεια βρίσκεται ακόμη σε προκαταρτικό στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να <clears throat> στοιχειωτηθεί η παράβιαση τη Οδηγία 85-337 ΕΟΚ και κατά συνέπεια τη Οδηγία 99-31 για τα απόλυτα. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται στην παρούσα φάσα παραβίαση τη κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα πολύ στενά. Ευχαριστώ ε, Υπάρχουν σχόλια. Φυσικά και την κρατήσουμε ανοιχτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αναφορά 24. Α, σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Σας παρακαλώ. Ε, όχι, καθίστε. Αν αισθάνεστε καλύτερα, αν αισθάνεστε άνετα, δεν χρειάζεται να σηκωθείτε. Ωραία, ό,τι θέλετε. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέταξε την αναφορά μου στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον σας και την προσήλωσή σας στα ιδεώδη ε, των πατέρων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήθελαν μια Ευρώπη χωρίς ε, σύνορα μετά από τις συγκρούσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών που παρά ε, τα πολλά της καθήκοντα ε, κατέβαλε ε, πολλές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αναφοράς μου και επέδειξε ιδιαίτερη επιμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων της. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενδιαφέρθηκαν για την αναφορά μου και μα υποστήριξαν. Η Επιτροπή Αναφορών σήμερα μου δίνει την ευκαιρία να σα να συμμεταφέρω την άποψη ε, των πολλών φαρμακοποιών που ε, ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν μπορούν, ε, δεν μπορούν, δεν αναγνωρίζεται το, το επαγγελμά του Με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται ως παρείε, ως φαρμακοποιοί δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, ένας βρετανικό νόμος του απαγορεύει σε κάθε Ευρωπαίο ε, φαρμακοποιό που δεν πήρε το πτυχίο του σε ε, πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου να εργαστεί ε, ω υπεύθυνο φαρμακοποιό σε ένα καινούριο φαρμακείο με διάρκεια. Όταν, όταν έχει, το, φαρμακο, το φαρμακείο αυτό έχει ξεκινήσει πριν από λιγότερο από τρία χρόνια. Αναχρονιστική λοιπόν αυτή η απαγόρευση και πρέπει να σας πω ότι απαγορεύεται η δημιουργία νέων φαρμακείων. Παρά το γεγονός ότι έχουν γραφεί ε, στο Φαρμακευτικό Σύλλογο εδώ και πολύ ε, καιρό. Και ανεξάρτητα με την επαγγελματική εμπειρία του συγκεκριμένου προσώπου. Συγκεκριμένα, αυτό τι σημαίνει. Ότι ένας Ευρωπαίος φαρμακοποιός, ο οποίος σήμερα ε, κρατάει ένα φαρμακείο στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 10 χρόνια, θα ε, πάυσει να ασκεί την δραστηριότητά του εάν μεταφέρει το φαρμακείο του 100 μέτρα ε, πιο κάτω. Να σας μιλήσω για την ιστορία μου. Την ιστορία ενός καθημερινού Ευρωπαίου πολίτη ο οποίο το 1998, μετά από τρία χρόνια στο Ταμείο Ανεργία στη Γαλλία, με γυναίκα και τρία παιδιά, ε, σήμερα βεβαίως, είμαι πατέρας 14 παιδιών, μετέφερα ε, τη δραστηριότητά μου στο Ηνωμένο ε, και ε, το 1998 με μεγάλη μου έκπληση ανέλαβα ένα φαρμακείο μιας αλυσίδας. Και με βάση τον, την, με, με, βάση την, τον νόμο της ε, Γαλλίας αναφερόμουν ε, ως παράδειγμα ε, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 1999 έγινα ελεύθερος επαγγελματίας και βρέθηκα απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα του, ε, αυτής της νομοθεσίας που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις, στις 11 Μαΐου του 2007 ενημερώθηκα για το γεγονός ότι το πτυχίο μου δεν μου επέτρεπε να αναλάβω ένα καινούριο φαρμακείο στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Και στις 30 Σεπτεμβρίου του 2008 ε, ε, με αντιμετώπισαν ως κοινό εγκληματία αν θέλετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και ε, ε, πλέον δεν μπορούσα καθόλου να συμμετέχω σε αυτά τα φαρμακεία, στα Άσδα. Έγινε προσφυγή στο Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και πιστεύω ότι ε, δίδεται διακριτική μεταχείριση ε, του αυτού του απαρχιωμένου, του παροχημένου νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια προσέφυγα στον Νότιο Δικαστήριο ε, και ζήτησα και αποζημίωση ταυτόχρονα και ενδεχομένως και προδικαστική ερώτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να ερμηνευτεί το βάσιμο του συγκεκριμένου νόμου με τη συνθήκη. Και εδώ δεν είχα ε, επιτυχία όμω, διότι το Ανώτατο Δικαστήριο στι 14 Οκτωβρίου 2009 θεώρησε ότι το ΕΒ δεν παραβιάζει καμία διάταξη του κοινοτικού δικαίου και δεν είχε νόημα υποβολή προδικαστική ερώτηση, διότι ήδη είχε γίνει η προδικαστική ερώτηση το 2005 από το Ανώτατο Δικαστήριο. Εγώ το αμφισβητώ βεβαίω, διότι το συγκεκριμένο ερώτημα ε, το οποίο είχε τεθεί τότε δεν είναι το ίδιο με αυτό το οποίο υπέβαλα εγώ στι 14 Οκτωβρίου 2009 λαμβάνοντας υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δηλαδή ε, την, ε, το, ε, το κατά πόσον κάποιος, κατά πόσον ευσταθεί ο νόμος αυτός απέναντι σε ένα άτομο το οποίο δούλευε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασκούσε το επάγγελμα πάνω από 10 χρόνια. Στις, τον Αύγουστο 2009 αλλά και τον Οκτώβριο του 2009 απευθύνθηκα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τότε μου, μου ζητήθηκε να υποβάλω το έτοιμά μου στην Επιτροπή Αναφορών γιατί εσείς τα αρμόδιοι. Γι' αυτό στις 14 Οκτωβρίου 2009 υπέθεσα κατέθεσα ε, προσφυγή ε, ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για παραβίαση καθηκόντων, για παραβίαση κοινωνική νομοθεσία, επειδή δεν δέχτηκε το Ηνωμένο Βασίλειο να υποβάλει προδικαστική ερώτηση. Νομίζω ότι ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε πει ότι ένα πολίτη που ζητά προδικαστική ερώτηση ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, εάν δεν ε, με βάση τα εκεί άρθρα τη συνθήκη, εάν δεν δοθεί συνέχεια στο αίτημά του όταν πρόκειται ε, για ένα, για ένα θέμα τέτοιο, έχει δύο επιλογέ. Να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με βάση του ε, συγκεκριμένου άρθρου τη συνθήκη μπορεί να συγκαλέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή να ασκήσει προσφυγή απευθεία στο συγκεκριμένο κράτο μέλο. Η δεύτερη όμω επιλογή δεν είναι δυνατή στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα τι μου απομένει η πρώτη επιλογή, που προφανώς είναι η βέλτιστη, γιατί προσφέρει την εγγύηση ισότιμης αντιμετώπισης. Πράγμα το οποίο προσφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί, ε, ε, ε μπορεί να εξεταστεί το ζήτημα του συγκεκριμένου πολίτη και ενδεχομένω ο πολίτη αυτό θα μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση συνέχεια. Όσον αφορά το αίτημά μου, η Επιτροπή με βάση παρατηρήσει συμπέρανε ότι. Ε, ότι λανθασμένα ερμηνεύεται από το Ηνωμένο Βασίλειο το συγκεκριμένο θέμα και από την άλλη ότι θα πρέπει το αίτημα, ε, του, ε, το, αίτημα το συγκεκριμένο θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση το άρθρο 43 της ε, συνθήκης και να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Το Ηνωμένο Βασίλειο στην απάντησή του επιμένει στην στην λαθασμένη ερμηνεία τη συγκεκριμένη οδηγίας. Η Επιτροπή λοιπόν στις παρατηρήσεις, στις συμπληρωματικές παρατηρήσεις ε, της ε, 22ης ε, ε, Ιανουαρίου του 2010 παραπέμπει στην ερμηνεία του 2009 και ανακοινώνει την πρόθεσή τη να έρθει εκ νέου σε επαφή με το Ηνωμένο Βασίλειο για να εξεταστεί η συμβατότητα των συγκεκριμένων διατάξεων με τη συνθήκη. Δεν ήρθε λοιπόν ο, ο καιρό η Επιτροπή να αντλήσει όλα τα συμπεράσματα ε, και να μην, να μην ε, ο πολίτη, ε, ο Ευρωπαίο πολίτη, να αισθάνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί στη μοίρα του. Παρά όλα αυτά τα οποία είπαν οι πατέρε ε, των συνθήκων το, 1957 στην Ρώμη. Και τι, και τι γίνεται με τι υλικέ αλλά και ηθικέ ζημίε που υπέστη. Ε, το, Κοιτάξτε, ε, πρέπει να σας πω ότι ε, παρά τις ε, προσφυγές που έχουν γίνει, αυτή τη στιγμή το μόνο που μου μένει είναι η συνέχεια που θα δοθεί στην αναφορά μου. Με βάση αυτά που υπέβαλα στις, τον Οκτώβριο 2009. Τελειώνω. Απευθύνω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσετε τα προνόμια σα με βάση τα άρθρα 226 και 230, ε, δεύτερο εδάφιο των συνθηκών, και να απευθύνετε στο, δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη ε, στα θύματα του, ε, αυτού του συγκεκριμένου νόμου του, του, του Ηνωμένου Βασιλείου και, ε, ε, και αναφέρομαι επίση και στην Οδηγία 2005-36 τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενσωμάτωση ε, στο, στην νομοθεσία. Ε, ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτω η Γαλλία, ζήτω και το Ηνωμένο Βασίλειο. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέιχοκ από την Επιτροπή. Σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε και την παρουσίαση ε, του επόμενου ζητήματος, γιατί φαίνεται ότι είναι παρόμοια τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι οι δύο αναφορές που έχουμε σήμερα ε, είναι παρόμοιες και αναφέρονται ακριβώς στο ίδιο θέμα. Έχουν την ίδια προβληματική. Άρα λοιπόν η απάντηση που θα δώσουμε ε, και στο συγκεκριμένο αυτό θέμα αφορά και τη δεύτερη αναφορά. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ε, συνετό να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες του θέματος. Παρουσίασε τόσο ενδελεχώς ο αναφέρον. Απλά και μόνο θα ήθελα να διευκρινίσω τα νομικά πλαίσια και κυρίως τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν οι Βρετανικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναφέρονται στο άρθρο 24, ε, παράγραφος 4 της Οδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων για να αρνηθούν ε, στους κατόχους τέτοιων διπλωμάτων ε, την διαχείριση και την, ε, νέων φαρμακείων στην ε, Αγγλία. Αυτό το άρθρο λοιπόν ε, της οδηγίας βρίσκεται στο τμήμα της οδηγίας που οργανώνει την αυτόματη αναγνώριση. Η παρέκκληση του συγκεκριμένου άρθρου θα πρέπει λοιπόν να ερμηνευθεί ως παρέκκληση στην αυτόματη αναγνώριση, το τονίζω ή εν λόγω παρέκκληση. Δεν μπορεί λοιπόν να ε, παρεκκλίνει από του άλλου μηχανισμού αναγνώριση ε, που προβλέπει η οδηγία και σίγουρα δεν μπορεί να περιορίσει ε, τα δικαιώματα των πολιτών όπω προβλέπονται αυτά από τη συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί λοιπόν ότι η συγκεκριμένη κατάσταση όπω την παρουσιάζει ο κύριο Τάγκα είναι ιδιαίτερα προβληματική και ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφέ με τι αρχές, Βρετανικέ Αρχέ και θα εξακολουθήσουμε να μελετάμε την περίπτωση και αν προκύψει ανάγκη σίγουρα θα επευθυνθούμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν ε, το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ε, εάν τώρα δούμε ότι δεν υπάρχει παραβίαση ε, του κοινοτικού δικαίου, θα αρχιθετήσουμε την υπόθεση. Αυτά θέλω να πω και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, πράγματι, είναι ιδιαίτερα λυπηρό όταν ακούμε αυτά τα οποία μας είπε ο αναφέρον. Πραγματικά, από την άποψη της Επιτροπής μας, εγώ δεν βλέπω γιατί περιμένουμε και δεν απευθυνόμαστε απευθεία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κοιτάξτε, ε, οι Βρετανικέ αρχέ δίνουν πάντα την ίδια απάντηση. Την ίδια απάντηση σα δώσουν και τώρα. Εγώ, κοιτάξτε, αυτό που υποδεικνύω, προτείνω είναι να μην περιμένουμε και να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ειλικρινά, σα λέω ότι εδώ έχουμε την ευρωπαϊκή αγορά που θέλουμε να λειτουργήσει σωστά. Δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα, δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λέμε στους νέους ακριβώς να πάνε να εργαστούν παντού στην Ευρώπη και να μην σταματούν στα σύνορα ενό κράτου μέλους και ακούμε τέτοιες περιπτώσεις, τι να σας πω. Και κάτι άλλο. Πίσω από τη μία αναγνώριση, τι βρίσκεται αυτή η περίπτωση του κυρίου, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, ε, πραγματικά υπέστη ζημία. Ε, ήταν ε, στην ανεργία, έχει μια οικογένεια να, να ζήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά με σοκάρει αυτό το θέμα. Και ειλικρινά ζητώ, ειλικρινά ζητώ να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθεί απευθεία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ο κύριος Μποσινάρου, θα ξεκινήσω λέγοντά σας ότι για μένα αυτό είναι μια σαφής περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για διακριτική μεταχείριση. Διακριτική μεταχείριση που στηρίζεται σε κάτι που έρχεται ε, σε αντίθεση με το ίδιο το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, ε, αγαθών και κεφαλαίων. Κάτι το οποίο ε, ε, το, το θέλει και το Λονδίνο, έτσι. Δεύτερον, Δεύτερο σχόλιο. Θυμάμαι ότι πριν από δύο χρόνια, όταν συζητούσαμε την αναφορά ενός μέλους του, ε, ε, ε ενός ισπανικού ομίλου ε, ο οποίος αθλητικού, ο οποίος είχε ε, εκφράσει συγκεκριμένα παράπονα εναντίον όχι τη νομοθεσία Ισπανική, αλλά εναντίον των Ισπανικών κανόνων, που απαγόρευε σε ένα Ισπανό προπονητή να γίνει μέλο ε, τη βασιλική λέσχη τζόκεϊ, επειδή δεν είχε, ε, δεν είχε αποκτήσει την κατάρτισή του στην Ισπανία, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τότε είχαμε προτείνει ότι η Ισπανία και πολύ σωστά θα πρέπει να υπακούει στου κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, και τώρα βλέπω δεν ισχύει το ίδιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν πρόκειται για ένα φαρμακοποιό, ο οποίο ε, έχει έρθει από την υπηρετική Ευρώπη για να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα, πρώτα απ' όλα πρόκειται για διακριτική μεταχείριση. Και η διακριτική μεταχείριση είναι κάτι που θα πρέπει να τιμωρείται. Έτσι δεν έχω από τίποτα άλλο. Δεύτερο σχόλιο. Καταλαβαίνω ένα από του λόγου για του οποίου Ε, δεν ε, ήταν εκτός ε, της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Γιατί αυτό αφορά και ανθρώπινα δικαιώματα, μην το ξεχνάμε. Και όμως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί αύριο ένας Βρετανός γιατρός δεν θα μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμά του στη Ρουμανία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία και τότε τι θα γίνει. Ε, τελικά η Ευρώπη, τι θα είναι η Ευρώπη, άμα δεν μπορεί κάποιο να ασκήσει το επάγγελμά του κάπου αλλού. Ε, εδώ μιλάμε για προστατευτισμό, για ε, προώθηση εθνικών αξιών και όχι ευρωπαϊκών αξιών εμπροκειμένου. Και πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένη αυτή η αντίδραση τη Επιτροπή. Και δεν νομίζω ότι η δέσμευση είναι αυτή που θα έπρεπε. Ε, όχι, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και πρέπει να υπάρξει αντίδραση με συνεπή τρόπο. Να, να περιμένουμε και άλλα τέσσερα χρόνια. Όπω στην περίπτωση με τι πέτσε. Και τότε μετά θα αντιδράσουν οι αρχέ ε, του Λονδίνου ε, και τελικά θα αλλάξουν κάποια στιγμή την νομοθεσία. Μα είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Και πρώτα απ' όλα το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία του και δεύτερον, τιμωρηθεί αυτή η περίπτωση διακριτική μεταχείριση να τιμωρηθεί με τον σωστό τρόπο. Γιατί αν και άλλε χώρε κάνουν το ίδιο, τότε μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Αν έχουμε μια μικρότερη χώρα, τότε θα την αναγκάσουμε να, να συμπεριφερθεί σωστά. Άρα τι κάνουμε, εδώ δεν την υποχρεώνουμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι απαράδεκτο και έχετε καθήκον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναρθώσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου για να είμαστε συγκεκριμένοι. σύμφωνα και με αυτά που πρότεινε η κυρία Γκρουνή, θα έπρεπε, θα πρέπει μάλλον, να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έτσι. Και εμείς θα αποστείλουμε πολύ αυστηρή επιστολή προς τις Βρετανικές Αρχές. Δεν ξέρω, στο Υπουργείο Παιδείας. Και θα ζητήσουμε εξηγήσει για άλλη μια φορά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστώ. We uh, Συνεχίζουμε με το 28. Α, το 25. Η κυρία Αγγέλικα Κόμετ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά του κυρίου Αμπέλα αναφέρεται στον τίτλο σπουδών του μηχανικού και η άσκηση του επαγγέλματος στη Μάλτα και του αντισταθμιστικού μέτρου. 1η Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου ε, ε, απάντησα η Κομισιόν επιμένει στη θέση της της 3 η Νοεμβρίου με μία εξαίρεση υπάρχει ένα στοιχείο στο αντισταθμιστικό μέτρο που ζήτησε διευκρίνηση η Κομισιόν από τις Μαλτέζικες Αρχές. Αυτό το στοιχείο του αντισταθμιστικού μέτρου είναι η, ε, η μια διατριβή που ζητήθηκε για ένα σχέδιο μηχανολογικό. Στις 18 Φεβρουαρίου ζητήθηκαν από την Κομισιόν ε, διευκρινήσεις από τις Μαλτέζικες Αρχές και τώρα είμαστε εν αναμονή των διευκρινήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο. Λοιπόν, είμαστε στην υπόθεση στην αναφορά 25. Στο σημείο 25. Υπάρχουν παρατηρήσεις από τα μέλη. Κλείνουμε δηλαδή την αναφορά. Yes, possibly this is going to be... Πιθανόν θα κλείσουμε το θέμα αυτό και πάμε στο σημείο 26. Αφορά θέματα υγείας. Ο κύριος Σέργιο Νιόλα. Ο κύριος Σμίτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Στη γραπτή μας ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει κάποια πράγματα εις ό,τι αφορά την διαφήμιση, την τηλεοπτική διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων, δημόσια διαφήμιση και στην τηλεόραση. Οι διαφημίσεις επιτρέπονται για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και αν γίνονται διαφημίσεις θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν, ότι θα πρέπει να διαβάζονται οι οδηγίες που εσωκλείονται πολύ προσεκτικά και να συμβουλεύονται και γιατρούς ή φαρμακοποιούς. Αφού ελάβαμε την αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στην Ιταλία, ήρθαμε σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές, επειδή οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται και η τήρησή τους να εποπτεύεται από τις εθνικές αρχές. Ζητήσαμε λοιπόν να μάθουμε πρώτον πώς εφαρμόζουν την, ευρωπαϊκή, σχετική ευρωπαϊκή διάταξη και πώς την επιβάλλουν. Μας έδωσαν στοιχεία σχετικά με την σχετική εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας και μας ενημέρωσαν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές φροντίζουν για την πρακτική εφαρμογή και μας έδωσαν αντίγραφο ε, ενό Υπουργικού Διατάγματος ή Απόφασης που θέτει το θέμα στις αρμόδιες αρχές στην Ιταλία εκ νέου και ε, τους ενημερώνει σχετικά με τις προϋποθέσεις ε, σχετικά με τις διαφημίσεις και πώς θα αντιμετωπίζονται οι διαφημίσεις που δεν ε, συνάδουν με τους κανόνες. Αποκομίσαμε λοιπόν την εντύπωση από την απάντηση των Ιταλικών αρχών ότι ε, εφαρμόζεται ε, κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεύτερον ότι επαρκή μέτρα λαμβάνονται για την διασφάλιση της εφαρμογής αυτών των διατάξεων και σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση στην Ιταλία. Αν σας κατάλαβα καλά, το, παρακολουθούν το θέμα οι τελικές αρχές ή όχι. Το θέμα της ε, δράσης ε, κάποιων, της ε, θέσπισης μέτρων ε, που θα παρακολουθούν το θέμα των παραβιάσεων των τηλεοπτικών διαφημίσεων και των σχετικών κανόνων ε, επαφιέται στις εθνικές αρχές. Και αυτή η δράση στηρίζεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει όμως η εφαρμογή των διατάξεων να γίνεται από τις ε, ε, εθνικές αρμόδιες αρχές και οι Ιταλικές αρχές μας διαβεβαίωσαν ότι ε, λαμβάνουν μέτρα για να παρακολουθούν κάθε μεμονωμένη περίπτωση ώστε να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι κανόνες. Χωρίς μικρόφωνο. Okay. Health in Italy. Η υγεία στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Η αναφορά είναι από Ιταλό υπήκο που εργάζεται στο δημόσιο τομέα και παραπονείται σχετικά με τους αυστηρότατους, όπως λέει, κανόνες που ισχύουν για ασθενείς που πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι ή να κάνουν ε, εξετάσεις. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι εδώ πρόκειται για διακριτική μεταχείριση και απαντήσαμε ήδη γραπτός στην αναφορά αυτή ε, το κοινοτικό κεκτημένο σε αυτό το τομέα των ε, διακρίσεων ε, αφορά αναπηρίες. Δεν υπάρχει δηλαδή έδαφος για να στηριχθεί αυτή η προσφυγή. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για την απασχόληση που καλύπτει θέματα διακριτικής μεταχείρισης γενικότερα στην απασχόληση με βάση την ηλικία, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία που να ε, αφορά την άδεια για λόγους ασθενείας και αν θα υπάρχει ελεγκτής που θα πρέπει να το ε, εξετάσει αυτό. Είναι θέμα επικουρικότητας και τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να ρυθμίζουν το θέμα ε, Εκείνα. Γι' αυτό απαντήσαμε και προσπαθήσαμε να το διευκρινίσουμε το θέμα ότι η οδηγία πλαίσιο καλύπτει μόνο αναπηρίες και δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες σε σχέση με το τι επιτρέπεται ή όχι στα κράτη-μέλη επί του προκειμένου. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν και το, ε, και κτημένο δεν υπησέρχεται σε αυτό το θέμα, οπότε δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Ναι, αλλά διαρωτώ με εάν θα μπορούσαμε να στείλουμε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων την αναφορά αυτή για να αποφασίσει εκείνη, γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Και προς ενημέρωσή τους. Γιατί να εξετάσουν το θέμα, να το διερευνήσουν, γιατί μπορεί να συνιστά ε, κάποιας μορφής κοινωνικό πρόβλημα, σπάνιο μεν, κοινωνικό δε. Εσείς, που εσείς αποφασίζετε βεβαίως, εγώ απλώς προεδρεύω. Κοιτάξτε, για μένα αυτές οι αρχές της επικουρικότητας είναι αυτές που είναι. Πρέπει να κλείσει ε, η αναφορά. Ειλικρινά δεν είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα πράγματα, τι να σας πω, τα ξέρω κι εγώ. Ε, και στη Γαλλία έχουμε τέτοια περιστατικά. Είναι παρόμοια τα πράγματα, αλλά για μένα πραγματικά ε, το θέμα είναι αρμοδιότητα του κράτου μέλου και δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Εγώ είμαι στην Επιτροπή αυτή, αλλά για μένα ε, πρέπει να κλείσει η αναφορά. <laughs> Εντάξει, πρέπει να πω ότι με πείσατε.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 Uh, Annex um, Αυτές είναι... Πρόκειται για αναφορές που συνήθως κλείνουν και πρόκειται να κλείσουν εκτός αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση από κάποιο μέλος. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούν να κλείσουν αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Οι λίγοι δηλαδή που παρέμειναν. Thanks,